Bien. Mesdames et messieurs, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε. Έχουμε ένα εκπρόσωπο τουλάχιστον αναπολιτική ομάδα. Οι καλύτεροι είναι παρόντες. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Ξεκινάμε τη συνάντησή μα. Δεχόμαστε σήμερα το πρωί τον στρατηγό Σέρεν, ο οποίος από τον Νοέμβριο είναι πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε επίσης ε, δεχθεί και τον προκάτοχό του που ήταν υπεύθυνο μέχρι τον Νοέμβριο του 2009. Στρατηγέ μου, είναι η πρώτη σας εμφάνιση εδώ. Είχαμε βέβαια κάποιες επαφές αρκετά ενδιαφέρουσες και σχετικά καρποφόρες μέχρι τώρα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι που είναι εδώ παρόντες θα σας θέσουν αρκετές ερωτήσεις. Είναι αλήθεια ότι η Στρατιωτική Επιτροπή παραμένει για πολλούς από εμά ένας θεσμός λίγο απόμακρος. Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι τρεις αποστολές, οι στρατιωτικές αποστολές οι οποίες διεξάγονται σε αυτή τη φάση στα πλαίσια της ΚΕΠΑ η Αταλάντα στα ανοιχτά της Σομαλίας και στον κόλπο του Άντεν, το Άλτεα στο Κωσυφοπέδιο, στη Βοσνία συγγνώμη, και η τελευταία αποστολή, η εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αστυνομικές αρχές και αρχές ασφαλείας της Σομαλίας, η οποία διεξάγεται στην Ουγκάντα. Σας δίνω αμέσως το λόγο, στρατηγέ ΣΕΡΕΝΑ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι βουλευτές. Είναι μια καλή ευκαιρία για μένα να σας συναντήσω, τα μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και να σας ενημερώσω για τη δράση της Επιτροπής μας. Είχατε ε, ενημερωθεί από τον προκάτοχό μου τον ε, Σεπτέμβριο του 2009 χθες η Στρατιωτική Επιτροπή με 27 εκπροσώπους είχε την τιμή να έχει σαν ε, ε, ομιλητή σε, μια, σε ένα γεύμα εργασίας ε, τον πρόεδρο αυτής εδώ της Επιτροπής και τον ευχαριστώ πολύ για μια ομιλία η οποία άνοιξε νέες προοπτικές στα πλαίσια της ανάπτυξης της ΚΕΠΑ και πολιτικής άμυνας. Η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είναι ένα μείζο νέο βήμα στην εξέλιξη της ΚΕΠΑ. Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει άμεσα όλες τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται της ΚΕΠΑ. Ο ρόλος της Στρατιωτικής Επιτροπής παραμένει, θα έλεγα, απαράλλαγος στα πλαίσια της νέας Επιτροπής, αλλά ο ρόλος αυτής της Επιτροπής θα επηρεαστεί αρκετά πέραν της κανονικής εργασίας που συνδέονται με τις ε, παρούσες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες της Επιτροπής μας φέτος ε, προσπαθούν, έχουν σαν στόχο να εφαρμόσουν τις συνέπειες της συνθήκης της Λισαβόνας και να αναπτύξουν ένα στρατηγικό πρόγραμμα, ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ε, θα μας δείξει ακριβώς την πορεία προς το μέλλον στα πλαίσια της νέας συνθήκης. Θα επιμείνω σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο της Στρατιωτικής Επιτροπής. Είναι βασικό σημείο για να συνεχιστεί ο διάλογος μας σήμερα και στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο συμβαδίζει πλήρως και με τη δική σας πολιτική βούληση. Πέραν αυτού θα κάνω και ορισμένα σχόλια σύντομα για τις συνεχιζόμενες ε, επιχειρήσεις είσαστε αρκετά ενημερωμένοι, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος και θα σταθώ κυρίως σε κάποιες ανησυχίες και σε κάποιες προοπτικές. Τέλος, στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης θα δώσω και κάποια προσωπικά σχόλια, θα κάνω και κάποια προσωπικά σχόλια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το θέμα της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας. Η δημιουργία της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεάσει τις στρατιωτικές δομές και η ΚΕΠΑ θα ενσωματωθεί στα πλαίσια της νέας αυτής υπηρεσίας. Μέχρι τώρα κάθε εναλλασσόμενη εξάμενη προεδρία έχει δώσει νέα όθηση στη διαδικασία ΚΕΠΑ. Η διαδικασία αυτή ήταν μια δυναμική διαδικασία και είχε βέβαια πάντα σαν στόχο την ολοκλήρωση των στόχων του εξαμήνου. Και αυτό μερικές φορές είχε φανεί πάρα πολύ μικρό σαν χρονική περίοδο. Η συνθήκη της Λισαβόνας στην ουσία θέτει την, τον έλεγχο της ΚΕΠΑ στα χέρια του του εκπροσώπου. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώνεται ε, και ο ρόλος και αυξάνεται ο ρόλος των συνοδευτικών σωμάτων γύρω από την ΚΕΠΑ και καθορίζεται μια νέα, θα έλεγα, αντιμετώπιση και προοπτική μακροπρόθεσμη πλέον. Ένα από τα πρώτα βήματα σαν νέος πρόεδρος ε, της Στρατιωτικής Επιτροπής ήταν να επανεξετάσω ε, το μέλλον των προτεραιοτήτων της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΚΕΠΑ συνειδητοποιώ ότι αυτό το πρώτο βήμα είναι ένα προληπτικό σε εισαγωγικά βήμα το οποίο ε, θα συνεχιστεί ε, θα έλεγα σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκομένους. Πάντως η Στρατιωτική Επιτροπή είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις βασιζόμενοι στις πολιτικές καθοδηγήσεις, 27 υπεύθυνοι στρατιωτικοί, τους οποίους συναντώ, και οι εκπρόσωποι της Στρατιωτικής Επιτροπής, οι οποίοι είναι κάποιοι από αυτούς σήμερα εδώ, έχουν υποβάλει τις δικές τους προτεραιότητες ε, για τη Στρατιωτική Επιτροπή. Μέσα της νέας συνθήκης και μέσω της ερμηνείας της νέας συνθήκης, καταλήξαμε σε 131 σε εισαγωγικά αποστολές Προφανές ε, δεν μπορεί κανείς να υιοθετήσει τόσες πολλές και να αναλάβει τόσες πολλές αποστολές. Γι' αυτό ε, συνεχίστηκε η συζήτηση και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο στρατηγικής επιτροπής και καταφέραμε να συμπτύξουμε τις 131 αποστολές σε 5 στρατηγικές πλέον αποστολές τις οποίες θα επανέλθω. Καθεμία από τις 5 αυτές υποστηρίζεται από ορισμένες κομβικές γράσεις 19 κομβικές δράσεις και αυτές οι κομβικές δράσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτεραιότητες για την προάσπιση των συμφερόντων και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να ερμηνεύσει λοιπόν κανείς την πολιτική βούληση των κρατών μελών. Και όταν οι πολιτικοί ε, μας λένε να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα, εμείς εφαρμόζουμε τις προτεραιότητες τις οποίες τα ίδια τα κράτη-μέλη έχουν καθορίσει. Και όταν ο αρχηγός του επιτελείου ή ένα κράτος μέλος λέγει γιατί το κάνουμε αυτό, τότε μπορούμε να επανέλθουμε στα προαποφασισμένα και να προσπαθήσουμε να βρούμε στα πλαίσια της στρατιωτικής συνεργασίας μια διαφορετική λύση. Οι πέντε βασικές προτεραιότητες είχαν συμφωνηθεί από τους 27 επιτελάρχες τον προηγούμενο μήνα. Όλοι συμφώνησαν και είναι θα έλεγα μια σωστή βάση για τις εργασίες της Επιτροπής μας τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμα αυτό θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση, καταρχάς δίσκατέτος, έτσι ώστε οι νέες εξελίξεις να αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα με σωστό τρόπο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουμε και ορισμένες προσαρμογές για την συνεχιζόμενη εφαρμογή της συνθήκης. Ας επανέλθω τώρα στο συγκεκριμένο περιεχόμενο του προγράμματος αυτού. Προσπαθήσαμε να το εκφράσουμε με πολύ συνοπτικό τρόπο, έτσι ώστε να καταστεί κατανοητό και σε επίπεδο επικοινωνίας. Η πρώτη από τις πέντε στρατιωτικές αυτές ε, στρατηγικές προτεραιότητες είναι να βελτιωθούν οι επιχειρήσεις και η διεξαγωγή των επιχειρήσεων της ΚΕΠΑ. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ο πυρήνας ε, της προσπάθειας που κάνουμε. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα φόρα και τους μηχανισμούς που υπάρχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιστοποιήσουμε όλες τις αναφαινόμενες ευκαιρίες. Δεύτερον, να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη μιας συνολικής αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα βασικό μήνυμα στα πλαίσια της νέας συνθήκης είναι μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αυτό δεν είναι εύκολο. Σε συνεργασία με τους υπολείπους εμπλεκομένους στη Στρατιωτική Επιτροπή, προσπαθούμε να παίξουμε το ρόλο μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο ξεπερνά τη στρατιωτική μας, θα έλεγα, παρουσία, και έχει σχέση με την επίτευξη των στόχων της συνθήκης της Λισαβόνας για την συνολικότερη βελτίωση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολιτικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο συνεργειών ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Δημιουργούμε ένα νέο τοπίο. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για όλους μας έτσι ώστε αυτή η συνένεση που υπάρχει για μια πιο συνολική αντιμετώπιση να μπορεί να γίνει εφαρμοστέα το ταχύτερο δυνατόν. Και αυτή είναι λοιπόν μία από τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Η τρίτη στρατηγική προτεραιότητα είναι το να, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ε, επιχειρησιακές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Τα μαθήματα τα οποία έχουμε πάρει από τις αποστολές μας και από τις άλλες δραστηριότητες μέχρι τώρα ε, νομίζω μας βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε από κοντά τα μαθήματα των κρατών μελών έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή ε, θα έλεγα διεξαγωγή των προσπαθειών μας. πρέπει να συνεργαστούμε με διάφορες χώρες έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε τους εξοπλισμούς τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας για να καλύψουμε τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν. Και θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε και στον τομέα του εξοπλισμού. Σε σχέση με την ανάπτυξη των ικανοτήτων μας, η Επιτροπή ε, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και η σχέση αυτή βελτιώνεται σε μόνιμη βάση και θα επανέλθω σε αυτό. Η τέταρτη στρατηγική προτεραιότητα είναι το να συνεισφέρουμε στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο στρατιωτικός ρόλος μέσα σε ένα νέο πλαίσιο και ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει αρκετές προτεραιότητες όπως συνεργασία σε επίπεδο μονίμων δομών, αμοιβαία βοήθεια και τη ρήτρα αλληλεγγύης. Στα πλαίσια της εφαρμογής της συνθήκης και εφόσον αυτή καθορίζεται σαν στρατηγική προτεραιότητα, έχω την αίσθηση ότι την προτεραιότητα αυτή μέσα σε λίγο καιρό θα έχουμε εφαρμόσει τις φιλοδοξίες μας και θα έχουμε ολοκληρώσει αν θέλετε τον στόχο αυτό. Και η πέμπτη και τελευταία στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης σε επίπεδο στρατηγικής με οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση όπως επίσης και με τρίτες χώρες. Η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ είναι πάντα ένα θέμα το οποίο έρχεται σε συζήτηση. Οι δύο οργανώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Και τα Ηνωμένα Έθνη είναι σημαντικός μας εταίρος. Ο, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Αποστολές του ΟΗΕ ήταν παρόν στις τελευταίες μας συναντήσεις. Εγώ στα πλαίσια της σύντομης χρονικής περίοδου που έχω αναλάβει τις ευθύνες μου έχω ε, συναντήσει αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Ρωσία. Επίσης έχω προγραμματίσει επισκέψεις στη Μόσχα, στο Κίεβο και σε άλλες χώρες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή της πέμπτης στρατηγική προτεραιότητα, θα αναπτύσσουμε τις εταιρικέ στρατηγικέ σχέσει τι οποίες έχουμε, οι οποίες είναι σημαντικότατες μακροπρόθεσμα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν προσπαθούμε ε, να βελτιώσουμε τις παρεμβάσεις μας, τις επιχειρήσεις μας, συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων, κάλυψη των κενών σε επίπεδο μέσων και εξοπλισμών και ανάπτυξη των ε, εταιρικών στρατηγικών σχέσεων. Αυτή είναι η τομή στους οποίους επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Συγκεκριμενοποιούνται αυτές ε, οι δράσεις σε σχέση με τους στόχους και, τα και τις χρονικές προθεσμίες που έχουμε καθορίσει. Υπάρχουν μακροπρόθεσμες προτεραιότητες αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε κάποιο έδαφος, θα έλεγα, και βραχυπρόθεσμα για να διευκολύνουμε τα πράγματα και προσπαθούμε να λειτουργούμε με έξυπνο τρόπο και με ε, μειωμένο ε, αποτελεσματικότερα δηλαδή ε, σε επίπεδο κόστους. Παράδειγμα, έχουμε συναντήσεις της Επιτροπής σε εβδομαδιαία βάση και έχουμε και φυσικά μια ημερήσια διάταξη η οποία καθορίζεται και παρουσιάζεται μια εβδομάδα πριν τη συνάντηση και κάθε ένα από τα θέματα συνδέεται πάντα με μία από τις προτεραιότητες τις οποίες προανέφερα, έτσι ώστε πάντα γνωρίζουμε ότι κάνουμε κάποια θετικά βήματα. Και είμαι πάρα πολύ διστακτικός να δεχτώ θέματα προσυζήτηση τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, τις πέντε. Προσπαθούμε να είμαστε ιδιαίτερα επαγγελματικοί στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Τώρα για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται. Η εκτέλεση της των επιχειρήσεων και των αποστολών της ΚΕΠΑ είναι φυσικά η κυρίαρχη προτεραιότητά μας. Είναι το ορατό θα έλεγα αποτέλεσμα των συλλογικών μας προσπαθειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε δύο στρατηγικές επιχειρήσεις, τις οποίες ανέφερε ο πρόεδρος, και μία στρατιωτική επιχείρηση εκπαιδευτικού τύπου, δηλαδή Αταλάντη, Αλτέα και έχουμε ξεκινήσει και την εκπαιδευτική μας δράση στην Ουγκάντα. Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω και θα ξεκινήσω με την Αλτέα στην Βοσνία Ευζεγοβίνη η οποία είναι επιτυχής. Ξεκίνησε εδώ και έξι χρόνια μετά από την επιχείρηση S4 του ΝΑΤΟ και μετά από τις συμφωνίες του Βερολίνου Το Αλτέα ξεκίνησε με 7.500 άτομα προσωπικό άνδρες και γυναίκες και ο αριθμός προσαρμόζεται συνεχώς στην βελτιούμενη κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας και σήμερα μιλάμε για 2.000 άτομα. Η πολιτική κατάσταση στην Βοσνία παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη και η περαιτέρω εξαιρήσεις της στρατιωτικής αυτής παρέμβασης θα εξαρτηθεί τελικά από τις πολιτικές εξελίξεις και την πολιτική ε, λύση που θα βρεθεί στα θέματα αυτά ήδη από το καλοκαίρι. Σημερίζομαι τις ανησυχίες του στρατηγού Μακόλ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική εντολή όμως να συνοδεύεται πάντα και από τις απαιτούμενες δυνάμεις. Και έχουμε προχωρήσει ε, και έχουμε κάνει προτάσεις για το πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση μετά από τις εκλογές ε, του Νοεμβρίου για την καταπολέμηση της πειρατείας ε, στα ανοιχτά της Σομαλίας, Αταλάντα. Ξεκινήσαμε το Δεκέμβριο του 2008. Είναι η πρώτη ναυτική αποστολή και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της ΚΕΠΑ. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει σε μια γενικότερη διεθνή προσπάθεια με πλοία και αεροσκάφη από το ΝΑΤΟ, από την Ένωση των Ναυτικών Δυνάμεων και από μεμονωμένα κράτη. Οι διοικητές της Αταλάντα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την συλλογική διεθνή συμφωνία. Η αποστολή Αταλάντα είναι υπόδειγμα θα έλεγα για αποτελεσματική συνεργασία με δυνάμεις από άλλα κράτη. Έχει βρει πραγματιστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και σταδιακές λύσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας. 1,5 χρόνο λειτουργεί, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονική περίοδος και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παρά με τις επιτυχίες που έχουν οδηγήσει στην αποθάρρυνση κάποιων πειρατικών ενεργειών, η δράση στη θάλασσα δεν είναι θα έλεγα η καλύτερη λύση μακροπρόθεσμα για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Η αποστολή αυτή είναι μια αποστολή ε, η οποία εμπλέκει θαλάσσιες δυνάμεις, η οποία προσπαθεί να φροντίσει τα συμπτώματα θα έλεγα περισσότερο παρά τις αιτίες των προβλημάτων. Μόνο αν υπάρξει λύση των προβλημάτων στην ίδια τη Σομαλία θα υπάρξει βελτίωση της κατάστασης. Θα πρέπει να συγχυστεί τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται η αποστολή αυτή. Έχουμε προσπαθήσει ε, να καλύψουμε τις ανάγκες μας ε, με τη βοήθεια των μεμονωμένων κρατών μελών Παρ' όλα αυτά ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός ε, είναι κάτι το απαραίτητο και θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα 27 κράτη-μέλη. Στα πλαίσια σαν παράδειγμα μιας διετούς προοπτικής θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τα ίδια τα κράτη-μέλη να δουν τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Να προσθέσω ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική παρουσιάζει πολλά θετικά χαρακτηριστικά γιατί θα καλύψει καλύτερα τις ανάγκες και αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ και όχι μόνο για την Αταλάντη. Μπορεί να υπάρξουν νέες πολιτικές συγκυρίες που να απαιτούν αλλαγές και φυσικά κάποιες ε, θα έλεγα κάποιοι αυτοχεδιασμοί οι οποίοι λύνουν τα προβλήματα μέχρι τώρα καλό θα είναι να μην υπάρχουν στο μέλλον. Εδώ και λίγους μήνες έχουμε ξεκινήσει και μια νέα προσπάθεια βοήθειας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία μιας δομής ασφαλείας αξιόπιστης στη Σομαλία. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνει κανείς η αδίποτε εκτίμηση. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν με μακροπρόθεσμο τρόπο την προσπάθεια σταθεροποίησης ε, της κατάστασης σε επίπεδο δημόσιας τάξης στη Σομαλία. Έχουν υπάρξει ήδη κάποιες αλλαγές, ενημερωθήκαμε τις τελευταίες εβδομάδες και η αποστολή αυτή υποστηρίζεται από τα περισσότερα κράτη-μέλη και αποστέλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η εκπαιδευτική δράση ε, θα μπορέσει να πετύχει η απόλυτη επιτυχία ε, θα εξαρτηθεί από την, από την δυνατότητα απορρόφησης και ενσωμάτωσης αυτών των εκπαιδευμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αστυνομικών Τμήματων και Δυνάμεων Ασφαλείας από τον Μηχανισμό Ασφαλείας στην ίδια τη χώρα. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τώρα κάνω κάποιες προσωπικές περισσότερο παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω ότι η ανάπτυξη και η επιτυχία της ΚΕΠΑ εξαρτάται από τις συλλογικέ προσπάθειες όλων των κρατών μελών. Η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε το μέσο αυτό και εξαρτάται τώρα από την βούληση και τις δυνατότητες των κρατών μελών και των σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν τη σωστή εξέλιξη των πραγμάτων. Η Στρατιωτική Επιτροπή παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό των δυνάμεων αυτών από τη μία έχουμε να κάνουμε με τα επίπεδα κατανόησης και διάθεσης των δυνατοτήτων που έχουν τα κράτη-μέλη για να εξυπηρετήσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και από την άλλη να εναρμονίσουμε τις μελλοντικέ ανάγκες των κρατών μελών καλύπτοντας πάντα τα ίδια αυτά συμφέροντα. Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις μπροστά στην ΚΕΠΑ, παγκοσμίου επίπεδου θα έλεγα, και η ανάγκη προσαρμογής των δυνάμεών μας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι δυνάμεις μας εμπλέκονται στην διαχείριση κρίσεων σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Έχουμε περιορισμένες δυνάμεις και δυνατότητες όμως και θα πρέπει να δούμε ότι θα προσμετρηθεί το ποσοστό επιτυχίας των προσπάθειών μας από το ποσοστό εμπλοκής μας ουσιαστικά. Το κόστος ανάπτυξης των δυνάμεων αυτών βέβαια σε επίπεδο εθνικών κρατών, μεμονωμένων κρατών, είναι πάρα πολύ υψηλό. Τους ζητάμε να το αναλάβουν αναγνωρίζοντας ότι έτσι θα υπάρξει δυνατότητα ανάληψης ακόμα μεγαλύτερων αποστολών και επιχειρήσεων στο μέλλον. Νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις στο μέλλον σταδιακά θα πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ευρωπαϊκές ικανότητες παρέμβασης που θα είναι καρπός των συλλογικών προσπαθειών μας που δεν θα είναι μία απλή θα έλεγα πρόσθεση όλων των δυνατοτήτων των κρατών μελών αλλά κάτι περισσότερο. Υπογράμμισα ότι σε επίπεδο θεσμικό η Στρατιωτική Επιτροπή και η Υπηρεσία Άμυνας ε, συνεργάζονται με στενό τρόπο Αλλά παρόλα αυτά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι η ανάληψη πολιτικής βούλησης από πλευράς των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά και η δική σας υποεπιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Οι δυνάμεις των κρατών μελών θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια αλλαγή της κατάστασης. Θα πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς μας, θα πρέπει να συνδυάσουμε τις εθνικές εξειδικευμένες ικανότητές μας, να εναρμονίσουμε τις απαιτήσει σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο εξοπλισμών. Όλες αυτές είναι δυνατότητες μεσοπρόθεσμα ιδιαίτερα εφικτές. Το να συνεχίσει κανείς απομονωμένο σε εθνικό επίπεδο να λειτουργεί είναι κάτι το οποίο δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Θεωρώ ότι η παρούσα οικονομική κρίση θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν ισχυρός καταλήτης για να υπάρξουν αλλαγές στο μέλλον. Σύμφωνα με τις εμπειρίες που είχα σαν επιτελάρχη στη χώρα μου, βλέπω ποιες είναι οι ανάγκες και βλέπω ποιες είναι οι δυνατότητες. Τώρα είμαι εκπρόσωπος του συλλογικού συμφέροντος των, επιτελαρχών, των επιτελείων συγγνώμη, των κρατών μελών. Και πράγματι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις κοινέ πολιτικές επιθυμίες των κρατών μελών. Έχουμε λοιπόν πολύ δύσκολη δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ στρατηγέ. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η συζήτηση. Υπάρχουν τρεις συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Εγώ θα έχω δύο ερωτήματα από πλευρά μου. Το πρώτο ερώτημα που βρίσκεται στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του, του προηγούμενου αξιώματος που είχατε στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η Σουηδία προχώρησε, έχει πολύ προχωρήσει στην ε, συγκρότηση των battle groups των μορίων χωρών. Η Σουηδική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το περασμένο εξάμεινο, είχε διατυπώσει την επιθυμία να ξαναδεί κατά πόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τακτικές ομάδες. Μέχρι τώρα δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιηθεί. Μιλήσαμε για μεγαλύτερη ευελιξία ανάπτυξη των δυνάμεων αυτών, να γίνουν πιο επιχειρησιακές και να υιοθετηθεί αυτό το δόγμα τη χρησιμοποιήση των battle groups. Τι συμβαίνει, ε, τώρα βρισκόμαστε στη Στρατιωτική Επιτροπή. Και το δεύτερο ερώτημα. Μιλήσατε για μια εταιρική σχέση, μια σύμπραξη, κυρίω με του οργανισμού, φυσικά το ΝΑΤΟ, την Αφρικανική Ένωση. Τι γίνεται με τις συνεργασίες, τις εταιρικέ σχέσεις για ορισμένα θέματα που θα πρέπει να είναι πιο δομικά ε, σε τρίτες χώρες, γιατί στις τρεις στρατιωτικές αποστολές που αναφέρατε, που βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή τρίτων χωρών και ε, για ορισμένες από αυτές δεν είναι μόνο συμβολική συμμετοχή. Αναφέρουμε στη Βοσνία για παράδειγμα, διότι μία από τις πιο σημαντικές μονάδες της αποστολής Αλτέα είναι η Τουρκία, η οποία καλείται να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, αν όχι και σημαντικότερος παράγον με τα πολιτικά θέματα που μπορεί να θίγονται. Η Ρωσία χτυπά την πόρτα θα έλεγα και εκείνη ζητά να υπάρξει μια συνεργασία για ε, τις αποστολές της ΚΕΠΑ. Οι ε, πρωτοβουλίε Μέρκελ με που δημιουργούν ορισμένα θέματα και όσον αφορά την Αταλάντα, την επιχείρηση Αταλάντα. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, ε, μεγάλες δυνάμεις οι οποίες για τις ναυτικές επιχειρήσεις θα ήθελαν να συνεργαστούν πιο ενεργά με εσά. Κίνα, Ινδία αλλά και Ρωσία. Πώς λοιπόν τα διαχειρίζεστε όλα αυτά σε επίπεδο στρατιωτικής επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πασκού. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα δρόμο χωρίς πολλά αγκάθια, με λιγότερα αγκάθια στο νέο σας αξίωμα, παρά το γεγονός ότι ξέρετε θα υπάρχουν δυσκολίες. Γνωρίζετε ότι παρουσιάζονται αυτές οι προτεραιότητες και τις ε, αντιδράσεις που υπάρχουν, νομίζω ότι κατορθώσατε να αποφύγετε, να καταστήσετε την εργασία της Επιτροπής σας ε, δέσμιο της πολιτικής βούλησης των μελών. Όσο πιο πολιτικό γίνεται το περιεχόμενο, τόσο πιο πολύ δέσμοι θα είσαστε ε, στην πολιτική ανάμεσα στα μέλη. Και βλέπω ότι κατορθώσατε να παραμείνετε μακριά από την πολιτική. Δεύτερον, συμφωνώ μαζί σας ότι η κρίση μπορεί να είναι καταλήτης, διότι μας υποχρεώνει να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας, τους πόρους μας. Και γνωρίζετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί όπως ακριβώς σχεδιάζεται. Και εμείς θα πρέπει να αναζητήσουμε και άλλες ευκαιρίες Δηλαδή να αναγκάσουμε σε κοινή δράση εκεί που η μεμενωμένη δράση δεν μπορεί να αναλυφθεί λόγω έλλειψη πόρων. Τώρα, έρχομαι στα ερωτήματά μου. Δύο ερωτήματα. Έχουμε ορισμένα προβλήματα. Ε, πώς, εξαρτάστε από τους πόρους του ΝΑΤΟ και συνεπώς ε, από την Συμφωνία Βερολίνο-ΣΥΝ αυτή η κατάσταση ε, που δεν, που δεν θα μπορεί να, υλοποιηθεί το headline course. Το δεύτερο ερώτημά μου και ζητώ συγγνώμη για την αγνιά μου επ' αυτού. Σκέφτεστε ή σχεδιάζετε μια στρατιωτική εκπροσώπηση μέσα στις αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο εξωτερικό. Επειδή εδώ στις Βρυξέλλες έχουμε εκπροσώπους, στρατιωτικούς εκπροσώπους, υψηλόβαθμους, σε ορισμένες αποστολές των χωρών οι οποίες ενδιαφέρονται. Συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you, President. I would like to stand on a couple of points. We Πολύ. Μας παρουσιάσατε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Θα ήθελα να ζητήσω το εξή. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει δική μνήμα στη συνθήκη της Λισαβόνας ως προς τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και ε, ε, τον είπα το εξπρόσωπο, αυτή η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι θα υπάρχει τώρα ένας καλύτερος τρόπος ώστε να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Στρατηγικής Επιτροπής για τις μελλοντικές δράσεις. Δεύτερο ερώτημα για την πειρατεία. Υπάρχει ε, με συχνότητα αυτών των επεισοδίων στις ακτές, ε, στις ε, Σομαλίες και τι γίνεται με την αποστολή Αταλάντα. Τρίτο ερώτημα. Αυτό που ζήτησε ο συνάδελφος Πάσκου. Πώς η οικονομική κρίση γίνεται σχητή από τη Στρατηγική Επιτροπή υπό την έννοια ότι υπάρχουν περικοπές στον προπολογισμό και θα επηρεάσουν σίγουρα τους αμυντικούς προπολογισμού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Merci, Madame Ευχαριστώ, κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποια ερωτήματα για τους διάφορους τομείς επέμβασης. Καταρχήν το πρώτο έχει να κάνει με το Κονγκό. Οι αποστολές Γιούλαξ ε, και Αταλάντα από, ε, πριν από το, ξεκίνησαν πριν από, το, από την ε, Γιούπολ και παρατάθηκαν για 1,5 με 2 χρόνια. Η αποστολή πάλι για το Κογκό παρατάθηκε μόλις για 3 μήνες. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς ε, έγινε και γιατί είναι τόσο σύντομη αυτή η παράταση για το Κονγκό. Υπήρχε κάποια διαφορά, ας πούμε, για την διάρκεια της συνολική της επέμβασης και αν ναι, Ποια ήταν η διαφορά, ποιο ήταν το σημείο το ακαθόδες για την Αταλάντα. Ε, πρόσφατα αποφασίστηκε ότι ε, θα συνεχίσουν οι επεμβάσεις ε, και στον Νότο και, στην και στα Ανατολικά. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ως πού θα φτάσουν αυτές οι επεμβάσεις και επίσης θα φτάσουν μέχρι την ζώνη των 12 μιλίων οι επεμβάσεις αυτές και κατά την άποψή σας η... καλύπτεται η εντολή από τον ΟΗΕ και για τη Σομαλία. Στις 16 Ιουνίου δημοσιεύθηκε από τους New York Times μια έκθεση από, τους, από τον ΟΗΕ που λέει ότι είναι η κυβέρνηση της Σομαλίας μία από τους, ε, πιο, από τους μεγαλύτερους ε, ε, από τις κυβερνήσεις που παραβιάζουν τις αρχές του ΟΗΕ για το ότι χρησιμοποιούν παιδιά ως στρατιώτες. η Ευρωπαϊκή Ένωση τι προτίθεται να κάνει. Μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σε επίπεδο OTM παιδιά στρατιώτες. Μήπως πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς γίνεται. Και αν δεν υπάρχουν ας πούμε δεδομένα για την, για την ημερομηνία γέννησης αυτών των παιδιών ή τέτοιου είδους στοιχεία, πώς ακριβώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον στρατηγό Σέρεν για την παρουσία του. Συνεχίζει ένα διάλογο σε σημαντικό επίπεδο ανάμεσα στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ένωσης και το Κοινοβούλιο μας, το οποίο όπως ο στρατηγός γνωρίζει υποστηρίζει ιδιαιτέρως την ανάπτυξη της ΚΕΠΑ και έχει αποδείξει, έχει εγκρίνει μάλλον με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος μας ο κ. Νοζόν. Για μας οι προτεραιότητες τις οποίες αναφέρατε είναι δικές μας προτεραιότητες και θα βοηθήσουν στην δημιουργία, θα έλεγα, μιας διαδικασίας που θα μας οδηγήσει με τη σειρά της σε μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Κάποια ερωτήματα που έχω και που έχουν σχέση με αυτά τα οποία εσείς είπατε. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καταρχάς, όπως βλέπετε, η δομή συγκεκριμένη, η οποία έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά για τη διαχείριση των κρίσεων επίσης, και οι σχέσεις ανάμεσα στις συνιστώσεις αυτής της νέας δομής, και εδώ έρχεται το στρατιωτικό προσωπικό, η ΚΕΠΑ, η υπηρεσία άμυνας και οι οριζόντιες σχέσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτές, όπως επίσης και οι κάθετες μορφές συνεργασίας, ειδικά δηλαδή οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και μένει να καλυφθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει αυτά τα οποία μπορούσε για να διευκρινιστούν κάποιες πλευρές αυτής της περίπλοκης εξίσωσης λειτουργίας της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Σχετικά με αυτό που ονομάσατε Comprehensive Approach, είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε με αποτελεσματικότητα, είναι κάτι το οποίο συνδέεται επίσης με το θέμα των ελλείψεων σε επίπεδο δυνάμεων πόρων και εξοπλισμού. Πώς μπορούμε να δούμε σήμερα μια διαδικασία ενίσχυσης της συνέργειας ανάμεσα στην πολιτική διάσταση και τη στρατιωτική διάσταση διαχείρισης κρίσεων. Τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι πολλαπλά και δεν ξεχωρίζουν εύκολα μερικές φορές ο στρατιωτικός κλάδος από το πολιτικό κλάδο παρέμβασης. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον τη συνεργασία ανάμεσα στους δύο τομείς. Και με ποιο τρόπο μπορούμε να αναλάβουμε κοινέ δράσεις και να τις διαχειριστούμε είτε πολιτικά είτε στρατιωτικά, εκμεταλλευόμενοι το σύνολο των συνεργειών που είναι διαθέσιμες, παρά τις σημαντικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες χώρες, ιδιαίτερα στον δημοσιονομικό τομέα. Πάντα για τα δημοσιονομικά για τον προϋπολογισμό. Είναι απαραίτητη να υπάρξει η λειτουργία του λεγόμενου Ταμείου Εκκίνησης, το Startup Fund. για τις μόνιμες διαφρατικές συνεργασίες. Ποια είναι η δική σας άποψη του δικού σας οργανισμού θα πρέπει να επικρατήσει η αντίληψη της συμπερίληψης και της συνοχής και της γρήγορης εκκίνησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και στο τέλος δύο θέματα τα οποία ήδη συζητήσαμε χτες στα πλαίσια της στρατηγικής αντίληψης του ΝΑΤΟ και αφορά την πέμπτη δική σας προτεραιότητα. Το θέμα της συμπληρωματικότητας δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΝΑΤΟ. Υπάρχουν κάποια διφορούμενα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο έγγραφο της κυρίας Όλμπραϊτ, της ομάδας Όλμπραϊτ, σχετικά με τις δυνατότητες συνεργασίας και με την πολιτική διάσταση του ΝΑΤΟ. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη αυτής της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στην Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω με τα δύο ερωτήματα του Πρόεδρου. Το πρώτο σχετικά με το battle group, τις ομάδες μάχης των σκανδιναβικών χωρών, των βορείων χωρών. Το σημαντικότερο μέρος είναι οι επιχειρησιακές επιπτώσεις και είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε σχέση με την πολιτική βούληση. Έχουμε ολοκληρώσει τις πέντε αποστολές που ζητούνται από ένα battle group. Θα ήθελα να προσθέσω όμως το εξή ως εμπειρία μου, ότι αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο και για αλλαγή, για μετασχηματισμό. To think of we had, didn't have the, battle group in our και υπάρχει ε, αυτές οι ομάδες ε, ε, σχηματισμού μάχης υπάρχουν στο πρόγραμμά μας, διότι μας βοήθησε να αλλάξουμε το σύστημα διαχείρισης, να δούμε διαφορετικά τα συστήματα, να αλλάξουμε ε, τις προμήθειες, το σύστημα προμηθειών, να έχουμε μια ικανότητα και μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη, μας έδωσε διαφορετική σκοπιά για την ετοιμότητα και επίσης ένα νέο συνέστημα σχετικά με τις επιχειρήσεις. Δεν το θεωρώ λοιπόν ως επιχειρησιακό μέσο, αλλά και ως εργαλείο. Και το χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη για αυτό το σκοπό επίσης. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Στη Στρατιωτική Επιτροπή δεν υπάρχει κοινή αντιμετώπιση για το πώς να αλλάξουμε την αντίληψη. Η αντίληψη παραμένει. Υπάρχει όμως μια συζήτηση σχετικά με την ευελιξία και τη δυνατότητα χρήσης αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις για το πώς να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι σχηματισμοί μάχης ή μέρη αυτών ε, στις ανθρωπιστικές, στη μονάδα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, και έχω υπόψη μου την IT αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο είναι σαφές στην Επιτροπή είναι ότι οπωσδήποτε πάντοτε πρέπει να προσαρμοζόμαστε ε, και να τροποποιούμε αυτή την αντίληψη. Προς το παρόν όμως δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αλλαγέ. αλλά η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Και η προηγούμενη Προεδρία και η παρούσα Προεδρία συζήτησαν αυτό το θέμα για μακρόν. Επίσης, συζητήσαμε σε συντομία τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μέρη αυτών των ε, σχηματισμών μάχης ε, στην επιχείρηση Αλτέα εφεδρικά. Προς το παρόν όμως αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ευελιξία στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το δεύτερο ερώτημα, σχετικά με αυτή τη συνεργασία, τις εταιρικές σχέσεις, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα μεμονωμένα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εξακολουθούν να λειτουργούν μόνα τους. Πρέπει να δημιουργήσουμε συνεργασίες, εταιρικέ σχέσεις. Η μία από τις πιο σημαντικές συμπράξεις πρέπει να ξεκινήσει μέσα την, ε, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αργότερα θα σας μιλήσω για την Αφρικανική Ένωση, αλλά βλέπω ότι δημιουργούνται ομάδες ε, φύλακες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των σκανδιναβικών χωρών και την Ισλανδία και υπάρχει ένα μνημόνιο συνεννόησης εκεί. Ε, ε, δεν είναι μόνο λόγια. Υπάρχει συνεργασία για τις προμήθειες, για τις ασκήσεις, για την εκπαίδευση, για την συντήρηση και πολλά άλλα θέματα. Και αυτό δεν είναι κάτι το δαπανηρό και έχει αποτελέσματα από επιχειρησιακή άποψη. Επίσης, χθες πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία μεταξύ τεσσάρων χωρών ε, της ε, ομάδας Visegrad στην, Ευρωπαϊκή, στην Κεντρική Ευρώπη. Και επίσης υπάρχουν πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, παρόλο ότι ορισμένα δεν είναι ε, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει βούληση να δημιουργηθούν συνεργασίες για να ε, υπάρχει συντονισμός, ε, τα πράγματα είναι πιο αποτελεσματικά και φθηνότερα. Τώρα, για τις τρίτες χώρες. Ε, συζητήσαμε για μακρόν στην Επιτροπή αυτό το θέμα και είμαστε ευτυχείς που η Ουκρανία συμμετέχει στην επιχείρηση Αταλάντα. Παρόλο που έχουμε συζητήσεις με ε, τη Ρωσία και της άμυνας έχουν προσκληθεί για την επόμενη συνάντηση. Την τελευταία φορά είχαμε τον επιτελάρχη της Ουκρανίας και όπως είπα στην αρχή χτυπά την πόρτα μας η, Κινία, η Κίνα. Χθες συζήτησαμε την αντιπροσωπεία και μιλήσαμε ε, για την επιχείρηση στον Ειδικό Ωκεανό αλλά και για ορισμένες επιχειρήσεις ασκήσεων και εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλές μορφές συνεργασιών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους οργανισμούς και με τις τρίτες χώρες. Είτε κοντά βρίσκονται είτε μακριά. Το δεύτερο ερώτημα σχετικά ε, με την εξάρτηση από τους σπόρους του ΝΑΤΟ. Ε, μιλήσατε για, ως παράδειγμα για το Βερολίνο ΣΥΝ. Ε, στην επιχείρηση Αλτέα είδαμε ότι με τις ρυθμίσεις Βερολίνο ΣΥΝ ε, υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Τουρκία που θα συμβάλλουν σημαντικά σε αυτή την αποστολή. Και το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση όταν ε, Ε, δεν ξέρω αν η σωστή λέξη εδώ είναι εξάρτηση, αλλά κατά πόσον αυτή η σχέση υπάρχει με μια άλλη χώρα όπως η Τουρκία που δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν ορισμένα ειδικά στοιχεία τα οποία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, στα μέσα που διαθέτουμε. Και θα πρέπει να ανοίξουμε τότε την πόρτα στις τρίτες χώρες και να προτείνουμε τέτοιες συνεργασίες. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας σχετικά με την ενοποίηση του στρατιωτικού, το μη στρατιωτικού σκέλους και να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είμαι ο πρώτος που επιθυμεί να υπάρχει διαφάνεια μεταξύ του στρατιωτικού και πολιτικού σκέλους και καλούμε τους, τους στρατιωτικούς συνδέσμους ή τους συναδέλφους από τα μη στρατιωτικά ε, όργανα. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τι πιστεύουμε από πλευράς Επιτροπής. Ο προκάτοχός μου είχε ε, γράψει μια επιστολή πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία και ανέφερε ποιες είναι οι επιθυμίες μας. Συζήτησα με τους υπευθύνους και δεν μπορώ να έχω εγγύησεις βέβαια, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ο ρόλος μου ως στρατιωτικού συμβόλου στον ύπατο εκπρόσωπο ισχύει πάντοτε και ότι το στρατιωτικό επιτελείο ε, εκτελεί τις βασικές ενέργειες που υπάρχουν και είμαι συντονιστής για τα 27 κράτη-μέλη. Αυτά τα τρία θέματα λοιπόν τέθηκαν και από τον προκάτοχό μου και νομίζω ότι ακόμα ισχύουν. Η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Ασχολούμαι με την αναδιοργάνωση των εργασιών και προσωπικά δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα που έρχονται στη δουλειά μέσα τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη δουλειά μας. Και ε, έχουμε απλά ένα μέρος της λύσης. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα έτσι. Ε, αναμένω ε, την ε, έγκριση της πρότασης από το Κοινοβούλιο αρχές Ιουλίου. Εξ όσο γνωρίζω όμως, αυτά είναι τα τρία στοιχεία από ε, τα, οποία παρτίζουν τη Στρατιωτική Επιτροπή, δηλαδή οι συμβουλές τον είπατε πρόσωπο στο στρατιωτικό επιτελείο και στα κράτη-μέλη. παίρνω τις ερωτήσεις με τη σειρά. Τώρα, για την πειρατεία και τη Σομαλία. Νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Εξαρτάται και από τον καιρό, εξαρτάται από την απειλή, εξαρτάται από το παγκόσμιο πρόγραμμα επισητισμού. Υπάρχει μια ευελιξία. Ο μόνος περιορισμός μας είναι ότι κάποια από τα πλοία δεν είναι τα κατάλληλα για να τα έχουμε σε ανοιχτή θάλασσα για κάποιες συγκεκριμένες περιόδους, οπότε τα μετακινούμε προς τον κόλπο του Άντεν. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων που έχουμε και οι πόροι πάλι επίσης ποικίλουν ανάλογα και με τις συνθήκες τις ε, καιρικέ. Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα για την οικονομική κρίση. Το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή αυτό πολλές φορές. Όλοι ξέρουμε ότι πολλά κράτη-μέλη, σχεδόν όλα, εν πάση περιπτώσει, ε, έχουν μειώσει δραματικά τους προπολογισμού τους και το ερώτημα πάντα είναι ότι όταν δημιουργούμε μια τέτοια μεθοδολογία ποιος θα την αναλάβει, ποιος θα είναι ο καθοδηγητής γιατί πάντα πρέπει να, έχουμε, να υπάρχει πολιτική βούληση για να τον αναλάβει κάποιος. Προς το παρόν η οικονομία είναι αυτή που μας οδηγεί και οι αλλαγές που υπάρχουν όντως είναι σημαντικές. Κατανοώ ότι τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται πως ε, δεν αξίζει τον κόπο να παραπονούνται. Ε, απλώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούμε. Και νομίζω ότι αυτή η κρίση μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για την συγχώνευση των κρατών, για τη συνεργασία του και για την κοινή τους δράση. Και αυτό με φέρνει στο ερώτημα για την ε, μόνιμη ε, συνεργασία. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το τι ακριβώς είναι αυτή η μόνιμη συνεργασία διαρθρωτική συνεργασία. Η παρούσα Προεδρία έχει κάνει ένα σεμινάριο για το θέμα αυτό και ξέρω ότι η επερχόμενη Προεδρία επίσης θα πράξει κάτι ανάλογο. Ε, εγώ φοβούμαι ελαφρώς ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές από την αρχή, να μην μείνουμε στο θεωρητικό. Και δεν μιλώ για, την, για το σύνολο της Επιτροπής, αλλά τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές και να ξεκινήσουμε πρακτικά από την αρχή. Ας πούμε, τα, οι σχηματισμοί μάχης, ε, πρέπει, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Είναι ένα θέμα που εμπίπτει στα πλαίσια της συνεργασίας. Ε, οπότε ας βάλουμε αυτό ως βάση και μετά ας αρχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό και ας προσπαθήσουμε να δούμε πού μπορούμε να δράσουμε και πού μπορούμε να δράσουμε καλύτερα ε, στην συντήρηση, στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς. Μόνο μια ρεαλιστική προσέγγιση ε, θα μας βοηθήσει, συγκρίνοντας δηλαδή το, τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να προχωρήσουμε. Αν υπάρχει κάτι θετικό από αυτή την ε, οικονομική κρίση, είναι ακριβώς αυτό, ότι μπορεί να αποτελέσει τον καταλήτη για τη συνεργασία. Του λεχθέντος, ε, κατανοώ απόλυτα και το ότι έχουμε να κάνουμε με 27 κυρίαρχα κράτη. Φυσικά είναι θέμα πολιτικής βούλησης και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και στα διάφορα κρατημέλη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, φυσικά. Αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα, αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, νομίζω ότι θα φροντίσει για τα πάντα η μηταραφύση. Αυτό είναι απλά μαθηματικά για μένα τουλάχιστον. Και χωρίς καμία εδώ ε, ευαισθησία λέω ότι πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία τώρα και να δράσουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τα μαθηματικά έτσι λένε. Επιχειρήσεις. Επέκταση των αποστολών. Στην Δημοκρατία του Κονγκό είτε μέσω της Αταλάντα ε, βασιζόμαστε και πάλι σε πολιτικές αποφάσεις. Τώρα υπάρχει πολιτική βούληση να επεκταθούν οι επιχειρήσεις και γεωγραφικά και χρονικά. Η επιχείρηση Αταλάντα, ας πούμε, να φτάσει μέχρι τις ακτές της Σομαλίας. Και αυτό είναι μια προοπτική για δύο χρόνια. Στην, ε, στο Κογκό ήταν, ε, είχαμε μια προοπτική τριών μηνών, αλλά αυτό έχει να κάνει με την πολιτική βούληση και με το τι θέλει και το Κονγκό. Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω την ερώτηση για τα πιστοποιητικά. Δεν ξέρω τα συγκεκριμένα αυτά δεδομένα που ζητάτε. Μπορώ να επανέλθω, όμως θα προσπαθήσω να μάθω. Η κοινή πολιτική άμυνας και η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και πώς μπορούν να συνεργαστούν και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κρίση. Πάλι δεν μπορώ να σας ε, απαντήσω επακριβώ, αλλά σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι αυτή είναι η δεύτερη στρατηγική μας προτεραιότητα, οπότε ε, δίνουμε μεγάλη σημασία. Όταν η υπηρεσία ε, εξωτερικών δράσεων αρχίσει να λειτουργεί, θα αποτελέσει έναν οργανισμό που για πρώτη φορά συνδυάζει πολιτικές και στρατιωτικές, στρατιωτικά μέσα και αυτό είναι το νόημα. Είναι μια συνολική προσέγγιση. Μιλούμε για μια συνολική προσέγγιση εδώ και καιρό, αλλά τώρα, εφόσον θα ιδρυθεί αυτή η υπηρεσία, θα έχουμε αυτή τη δομή και θα μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές. Και μετά θα μπορούμε να ε, γκρεμίσουμε και τους ορατούς και τους αόρατους τείχους που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων αρχών. Αυτή είναι η δική μου ευθύνη στην Επιτροπή, να το συζητήσουμε πολύ ε, ανοιχτά και να είμαστε ρεαλιστές. Και είμαι πεπισμένος ότι θα επανέλθουμε στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ομάδες, ε, του σχηματισμούς μάχης, ε, το, όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Για την συνολική προσέγγιση τώρα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων, θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν έχουμε κοινή άποψη στην Επιτροπή ως προς αυτό, ε, γιατί ε, ε, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Αλλά αν τηρήσουμε τις αρχές εδώ, η συνολική προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων δεν είναι θέμα στρατιωτικό, δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι θέμα πολιτικής. Και εκεί υπάρχει τελείως διαφορετική οπτική. πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη στρατηγική από το ΝΑΤΟ για, το, για τα συστήματα ελέγχου. Αλλά αν το δούμε αυστηρά στρατιωτικά, το να έχουμε ένα κέντρο επιχειρήσεων στο οποίο να μπορούν να λειτουργήσουν οι στρατιωτικοί, φυσικά είναι καλοδεχούμενο. Αλλά πρέπει να γίνει, να μπει σε κάποιο πλαίσιο γιατί αυτό κοστίζει και με τους περιορισμένου πόρου που έχουμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το κατά πόσο θέλουμε να κτίσουμε ένα νέο κτίριο ας πούμε ή αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι ένα αναπόφευκτο, αλλά προς το παρόν είναι πολύ νωρί ακόμη και ακόμη δεν έχω και όλα τα κομμάτια του παζλ για να σα δώσω μια πλήρη απάντηση. και για την έναρξη του Ταμείου και αν θα υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ή αν θα είναι ο κανονισμός ε, ε, πιο αποτελεσματικός. Νομίζω ότι η ε, Στρατιωτική Επιτροπή Περισσότερο ανησυχεί όταν έχουμε να κάνουμε με στρατιωτικές διανέξει. Ε, οι στρατιωτικοί ούτως ή άλλως ε, δεν ασχολούνται με τα ε, νομισματικά. Αν εμείς μπορέσουμε να φέρουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και να διευκρινίσουμε ακόμη καλύτερα τα πράγματα, τότε αυτό φυσικό θα είναι καλό. Η Επιτροπή θα μπορέσει ίσως να το ακολουθήσει. Οπότε όντως χρειάζεται βελτίωση. Νομίζω απάντησα στα ερωτήματα. Λοιπόν, όσον αφορά τα πιστοποιητικά γεννήσεω για του Σομαλούς, Βεβαίω ε, πρέπει να το δούμε. Αν μου επιτρέπετε, είχα παρακολουθεί αυτό το θέμα ε, από πλευρά των γαλλικών δυνάμεων που είχαν συμμετάσχει ε, στο σχηματισμό ορισμένων ε, δυνάμεων ασφαλείας ε, της Σομαλίας. Υπήρχε ένα τρίγωνο, αν θέλετε, για την πιστοποίηση της ταυτότητας, διότι δεν υπήρχαν πιστοποιητικά γέννηση, ε, είτε ήταν ελλειπή. Είχε γίνει μια δουλειά με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, τη μεταβατική κυβέρνηση Σομαλίας και με την επιτόπου αποστολή της Σομαλίας και με ειδείς μέσεις για να δούμε ποια ήταν η ταυτότητα ε, δηλαδή για τα, τους εκπαιδευμένους στρατιώτες και είχαν πρόβλημα με την ταυτότητά τους. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ορισμένοι αποκλείστηκαν από τους σχηματισμούς επειδή υπήρχε διαφορά σχετικά με την ηλικία τους. Φαντάζομαι ότι η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται, αλλά πρέπει να το εξακριβώσουμε. Κυρία Λόζιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και θα ήταν πραγματικά τρομακτικό να εκπαιδεύονται από την Ευρώπη παιδιά για να γίνουν στρατιώτε. Ε, ε Όντω ήταν πολλά τα ερωτήματα που σα τέθηκαν και φυσικά είναι δύσκολο να απαντήσετε λεπτομερώ σε όλα. Γι' αυτό μια ερώτηση ακόμα. Αυτή η κατάσταση στο Κονγκό ε, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Είπατε ότι ήταν, ε, έτσι ήταν τα πράγματα, τρεις μήνες για το Κογκό, ε, πολύ σύντομη περίοδος όντως και είπατε ότι το αποτέλεσμα έχει να κάνει με πολιτική απόφαση, βούληση. Ωραία. Ποια ήταν αυτή η πολιτική απόφαση τελικά, δηλαδή ελήφθη από κάποιους μεμονωμένα, αξιολογήθηκε, υπήρξαν κάποιες προτεραιότητες, ήταν ε, από την αποστολή, υπήρξαν κάποια προβλήματα που ανάγκασαν να είναι τόσο σύντομη αυτή η περίοδος. Και είπατε επίσης ότι πρέπει να δούμε και τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση δηλαδή του Κονγκό δεν θέλει να παραμείνουμε εκεί για περισσότερο χρόνο. Ε, θα ήθελα έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Και άλλο ένα ερώτημα για την Αταλάντα. Κατάλαβα σωστά δεν θα υπάρχει ε, περαιτέρω επέκταση de facto, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο να επεκταθούμε στις 12, στα 12 μίλια, στη ζώνη των 12 μιλίων. Αυτό για να το καταλάβω εγώ, για να είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Το μόνο που μπορώ να πω σχετικά με τη Σομαλία είναι το εξή. Ενώ επιλέγουμε εκπαιδευόμενους για την αποστολή στην Ουγγάντα, ε, έγινε πολύ πολύ προσεκτική επιλογή και ειλικρινά, ειλικρινά δεν παίρνουμε παιδιά. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Είδα τα στοιχεία, είδα τις διαφορετικές φυλές από την Σομαλία που εκπροσωπούνται στην αποστολή και πιστεύω ότι πάνω από 20% αντιδρούν. Υπάρχει αντίδραση για το 20% επειδή δεν, είχα, δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ο λόγος για τον οποίο διστάζω να απαντήσω στο ερώτημά σας είναι επειδή δεν μπορώ να σας πω ε, αν έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά θέματα, αν έχω πιστεί από τον επικεφαλή τη επιχειρήσεως ότι εκείνοι οι οποίοι τους επιλέγουν ελέγχουν την ταυτότητά τους και ότι τα άτομα αυτά είναι αξιόπιστα. Τώρα για το Κονγκό. Και εδώ οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες, διότι δεν έχουμε αναπτύξει δυνάμεις αλλά εξαρτάται το χρονικό διάστημα και από την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να αποσύρει τις μονάδες από το Κονγκό. Και αυτή η απόφαση λαμβάνεται πάντοτε ε, σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Κονγκό. Αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε διάφορες χώρες, ναι. Προσωπικά ε, υπήρχε διαφορά απόψεων σχετικά με την αποστολή ε, μονάδων στο Σουδάν. Ε, ας πούμε δεν μας ήθελαν στον Ταφούρ. Άλλες χώρες πάλι ζητούν να κάνουμε κάτι και μας καλωσορίζουν όπως στο Τσάντ. Ανάλογα με τις χώρες μας βλέπουν διαφορετικά και οι αποφάσεις είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα πάλι για την Αταλάντα τώρα. Η γεωγραφική κάλυψη. Πού λειτουργούμε, πού επιχειρούμε. 60 ε, μοίρες ανατολικά. Διότι πρέπει να βρούμε τους πειρατές που διαφεύγουν πέρα από αυτή τη γραμμή δεν μπορούμε να τους κυνηγήσουμε. Γι' αυτό επεκτείναμε την εμβέλειά μας, την κάλυψή μας. Τώρα για τα 20 ναυτικά μίλια, και αυτό είναι τεχνικό ερώτημα. Θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός στην απάντησή μου, γι' αυτό ε, να μου επιτρέψετε να επανέλθω σε αυτό το θέμα όταν έχω πλήρη εικόνα. Από τεχνική άποψη το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Bien, mon général, merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το πλεονέκτημα ε, ε, όταν έχει κανείς εκπροσώπους από το στρατιωτικό τομέα είναι ότι τηρούνται τα χρονικά όρια. Ευχαριστώ πολύ για την κάλυψη των θεμάτων. Θα πρέπει να γίνει μια νέα διαβούλευση για δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά, δύο ομάδε θεμάτων. Το ένα είναι το επιχειρησιακό, όπως θα το ονόμαζα, με παρακολούθηση των στρατηγικών αποστολών της Ευρωπαϊκής και το άλλο που θα είναι πιο ενιολογικό κυρίως όσον αφορά ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας και την εφαρμογή της, θα πρέπει να προσαρμόσουμε ορισμένες ρήτρε τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ε, και ε, θα... οι εξωτερικές σχέσεις είναι η προτεραιότητα, αλλά όταν ολοκληρωθεί το έργο θα δούμε μαζί ποιο θα είναι το περιεχόμενο και οι επιπτώσεις των νέων διατάξεων, κυρίως αυτής της ρήτρας της αμοιβαίας συνδρομής. Ευχαριστώ στρατηγέ μου και στο επανειδήν. Ε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας με το δεύτερο σημείο στην εμερήσια διάταξη. Θα δούμε τώρα το θέμα της γεωργίας. Πριν από την παρέμβαση του Πρέρ Μπέρ, επικεφαλής αποστολής στη Γεωργία, ο οποίος σε μια ώρα περίπου θα μας μιλήσει, ε, έχουμε τον κύριο Πορφίτζε σήμερα, ο οποίος είναι βοηθός Γενικού Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στη Γεωργία και έχουμε μία αποστολή η οποία θα μεταβεί στη Γεωργία τον Ιούλιο. Μεταξύ μας επίσης βρίσκεται ο κ. Κρίστοφ Ιζέ, ο αντιπρόεδρός μας που θα είναι στην αφέ της ηγητής για το θέμα της Γεωργίας. Συνεπώς νομίζω ότι είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, αυτά τα μέσα που έχουμε για τη Γεωργία, για να ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο της Γεωργίας δηλαδή πώς βλέπει η Γεωργία την ανάπτυξη της αποστολής μας και επίσης μία αξιολόγηση από την άποψη της Γεωργίας για το που βρίσκεται η κατάσταση Πρωτού μεταβούν τα μέλη μας επιτόπου. Εκεί θα έχουν σίγουρα συναντήσεις που θα εστιάζονται κυρίως ε, στην αποστολή ΕΜ και στην, στην ανάπτυξή της, αλλά γενικά για την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση ασφάλειας στη Γεωργία. Γι' αυτό σας δίνω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για το... Γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της γεωργίας. Τέσσερα πραγματάκια θα ήθελα να θίξω σήμερα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσε προσωπικό και βοήθεια σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να διατηρηθεί η ευαίσθητη, εύθραυστη ειρήνη που υπάρχει στη χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι είναι στο πλευρό μας και μας υποστηρίζει. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου θα αναφέρω τέσσερα πράγματα. Καταρχήν ότι είναι, πολύ, είναι απαραίτητη βοήθειά σας ε, για την ε, ασφάλεια των πολιτών μας και για τη σταθερότητα. Ε, δεύτερο, η Ρωσία μπλοκάρει την πλήρη ε, εφαρμογή της εντολής. Το τρίτο είναι ότι υπάρχουν τρομακτικές συνέπειες επιτόπου γιατί όντως ε, μιλούμε για ε, άρνηση των δικαιωμάτων, περαιτέρω στρατιωτικές δυνάμεις, μόνιμες απειλές στην κυριαρχία της Γεωργίας και το τέταρτο που θέλω να πω είναι ότι είναι απαραίτητο όχι να, απλώς να επεκταθεί η αποστολή, αλλά να πιέσουμε περισσότερο τους Ρώσους για να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ε, κατεχόμενες περιοχές που τώρα δεν είναι δυνατό. Η αποστολή που ε, δημιουργήθηκε το 2008 για να ελέγχει την ε, εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας ήταν σημαντική για την ασφάλεια επιτόπου. Θεωρούμε ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Γεωργία είναι βασική προϋπόθεση για τις περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον. Η Ρωσία ε, εδώ και χρόνια βλέπει την παρουσία διεθνών οργανισμών των, ε, του, όπως ο ΑΣΕ και άλλοι ως ε, εμπόδιο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εμπόδιο στις στρατηγικές της επιδιώξεις. Μετά από τα γεγονότα το 2008 με τη Γεωργία, η Ρωσία χρησιμοποίησε το δικαίωμα βέτο που έχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και εκμεταλλεύτηκε την ε, συνένεση και το σχετικό κανονισμό, ε, μηχανισμό για να μπλοκάρει την ύπαρξη αυτών των ε, οργανισμών στην Γεωργία. Οπότε τώρα δεν υπάρχει κανένα διεθνή οργανισμό στη Γεωργία που να έχει πρόσβαση στι περιφέρειε αυτέ ή να, απλώς να υπάρχει για να παρατηρεί την κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει η αποστολή της Ευρωπαϊκής στη Γεωργία παρά την επιθυμία της Γεωργίας να υπάρχει ο ΆΣΑ και, ο ΙΕ στην επικράτειά της και με την υποστήριξη της, ε, σχεδόν όλες της διεθνούς κοινότητας η Ρωσία το έχει μπλοκάρει. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο σημαντικό ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει γιατί είναι η μόνη παρουσία επιτόπου πια την οποία, για την οποία η, Ευρωπαϊκή, η Ρωσία δεν έχει δύναμη βέτο. Οπότε είναι σημαντικό, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή ε, Αποστολή να παραμείνει εκεί έχει εντολή η αποστολή σα ε, με ε, ε, έλεγχο της, συμφωνίας, της εφαρμογής της συμφωνίας για τα, με τα έξι σημεία για την επικράτεια της, Ρωσίας, για την επικράτεια της και την περιοχή της Απχαζίας. Δυστυχώς όμως η ρωσική κυβέρνηση έχει μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια για πρόσβαση σε τέτοιες κατεχόμενες περιοχές. Παρά τα διάφορα ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, η κατοχή εξακολουθεί να υπάρχει σε 20% τη ε, επικράτειας της Γεωργίας από τη Ρωσία. Και αυτό αποτελεί μεγάλη παραβίαση των, ε, του Διεθνού δικαίου και των, ε, και διαφόρων μνημονίων που υπάρχουν. Πριν αυτό, δεν, αυτό επιδεινώθηκε μετά το 2008 Μιλούμε δηλαδή για πολλές περιοχές, μικρά χωριά, σε συγκεκριμένες περιφέρειες και κυρίως στην Αυχαζία, ε, στις οποίες παρατηρούνται αυτές οι παραβιάσεις. Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί δυστυχώς ε, εκτοπίστηκαν από τις περιοχές τους λόγω των δράσεων που ανέλαβε η Ρωσία, από το 2008 κυρίως. και εκτοπίστηκαν από πολλές ε, ε, περιφέρειες ε, και από την Απχαζία. Και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν έχουν δικαίωμα να πάνε πίσω στα σπίτια τους. Μιλούμε για περίπου 400.000 γεωργιανούς που δεν έχουν, και για γεωργιανούς αλλά και άλλους πολίτες που δεν έχουν δικαίωμα γιατί υπάρχουν και κάποιοι μια μειονότητα εστονών που δεν έχουν ε, δικαίωμα. Έλληνες που έμεναν ε, κατά τη διάρκεια του 90 στην Αυχαζία. Προς το παρόν, η παραβίαση αυτή ε, σημαίνει ότι υπάρχουν 10.000 ε, Ρώσοι στρατιωτικοί. Τώρα υπάρχουν 10.000 στρατιώτες στην, ε, Ρώσοι στην, στην Γεωργία. Οι κατοχικές δυνάμει έχουν ε, καταστρέψει πολλέ ε, περιοχέ στην ε, περιοχή του Σινβάλια, στην Νότια Οσετία και σε άλλα μέρη τη χώρα, ώστε να δημιουργήσουν χώρο για περισσότερε στρατιωτικές εγκαταστάσει. Ήδη κάποιε από τι εγκαταστάσεις αυτέ έχουν ολοκληρωθεί. Η ίδια κατάσταση επικρατεί στην Απχαζία. Είναι μια διαδικασία εν εξελίξη και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ε, η έλλειψη, ο πληθυσμός που μεταφέρεται, που φεύγει, ε, κυρίως από την περιοχή του ε, είναι, ε, αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Μιλούμε για 10.000 άτομα τα οποία έχουν παραμείνει εκεί, ενώ παλαιότερα ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αυτό αποτελεί συνέπεια των ρωσικών δράσεων. Και οι περιοχές αυτές αδειάζουν. Οπότε αλλάζει και η δημογραφική κατάσταση της ε, περιοχής, της περιοχής και φυσικά αυτό επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης και των όσων μπαίνουν εκεί τελικά. Το άλλο κομμάτι που μας ενσυχεί είναι ότι οι Ρώσοι έχουν μετατρέψει την, ε, μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στην Τυφλίδα σε μια στρατιωτική βάση. Μιλούμε δηλαδή για 40 χιλιόμετρα ε, μακριά από, το, από την Τυφλίδα βρίσκονται αυτές οι εγκαταστάσεις και είναι πάρα πολύ κοντά και στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει δύο μεγάλα τμήματα της Γεωργίας αλλά και αποτελεί ένα μεγάλο σημαντικό σύνδεσμο για τις μεταφορές και το εμπόριο που είναι πολύ σημαντικό τμήμα της ε, γεωργιανής οικονομίας. Οπότε η στρατηγική αυτή τοποθέτηση των, ε, στρατα, των ε, και, λόγω, ε, και επειδή αποτελούν και μια, ένα ψυχολογικό κριτήριο εκφοβισμού για να πιστεύει ο κόσμος ότι βρίσκεται υπομόνιμη η κατοχή είναι, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Πέρα από αυτό υπάρχουν και αρκετοί περιβαλλοντικά κριτήρια. Επειδή ακριβώ δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν η Ρωσία, έχει ε, ξεκινήσει η εξόρυξη διαφόρων υλικών, ε, ξύλου, άμμου, για να τα χρησιμοποιήσει ε, για δικούς της σκοπούς. Η Απχαζία λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί ως, κομμάτι, ως περιοχή εξόρυξης για υλικών για κατασκευές από τη Ρωσία. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί τεράστιες ζημιές στην περιοχή. Οι προσπάθειες της ε, ε, κυβέρνησης είναι συνεχείς για να υπάρξει σύνδεσμος μεταξύ των ε, διαφόρων κοινοτήτων της Γεωργίας. Οι ανθρωπιστικές συνέπειες επίσης είναι πολύ σημαντικές. Τα τείχη αυτά που δημιουργούνται δεν δίνουν το δικαίωμα στου πολίτε να ταξιδεύουν ελεύθερα, να μετακινούνται ελεύθερα στη χώρα του. Οι κατεχόμενε περιοχέ ε, γίνονται γκέτο, όπου οι άντρε και οι πολίτες, οι και γυναίκες ζουν σε αισχρέ συνθήκε. Υπάρχουν βεβαίω τρόποι με του οποίου θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι και να το κάνει ειρηνικά και νόμιμα. Την 1η Ιουνίου το Λιθουανικό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα, το οποίο ε, αξιολογεί τις δράσεις ε, της ε, Ρωσίας και τις θεωρεί επιθετικές και την ύπαρξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας στην Αυγαζία ως κατοχή. Εμείς σεβόμαστε την απόφαση αυτή και ελπίζουμε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν όπως την απόφαση της Λιθουανίας. Μιλούμε λοιπόν για μια παράνομη κατοχή ενός κυρίαρχου κράτους, κράτους του, στον 21ο αιώνα και αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο οι πολίτες της ε, Γεωργίας ε, εκτιμούν πάρα πολύ και η κυβέρνηση της βέβαια την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, ένα, σε μια περίοδο που η παροχή στήριξη δεν είναι πολύ προφανής και θέλουμε να διατηρήσουμε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον όπως αυτό που υπάρχει τώρα στην Γεωργία. Και να σας πω για ποιους λόγους είναι αυτό σημαντικό. Γιατί είναι σημαντική η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να σας δώσω και παραδείγματα. Καταρχήν, σε πολλές ε, περιόδους έχουν υπάρξει κάποιες ε, φήμες που λένε ότι η κυβέρνηση κάνει, ε, ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό, η ευρωπαϊκή αποστολή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει δράσει σε αρκετές περιπτώσεις, όταν γινόντουσαν δηλαδή τέτοιες δηλώσεις. Η Γεωργία δεν έχει να κρύψει τίποτα. Πρέπει όμω να σα πω, έχουμε, κάνει, έχουμε συνάψει δύο συγκεκριμένα μνημόνια, συμφωνίε με την αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που, που επιτρέπουν την πρόσβαση τη Ευρωπαϊκή Αποστολή στι γεωργιανέ στρατιωτικέ δυνάμει. Επίση, έχουμε πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των στρατιωτών τη γεωργία, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή αυτή και αυτό αποτελεί μεγάλο κομμάτι των όσων κάνουμε για να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αλλά όταν μιλούμε για τέτοια διαφάνεια από τη δική μας την πλευρά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ένα κομμάτι το οποίο δεν πληρείται επαρκώς ή σχεδόν καθόλου ή δεν είναι διαφανέ. Τι γίνεται δηλαδή από την άλλη μεριά. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε πρόσβαση στι ε, κατεχομενες περιοχες περιοχέ. Δεν υπάρχει ούτε καν ένα ελεγκτή που να μπορεί να περάσει από την άλλη πλευρά για, από τι αποστολέ τι ελεγκτικές. Και σύμφωνα με την συμφωνία αυτό αναφέρεται, αυτό αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει τέτοια πρόσβαση. Επίσης, πρέπει να πω ότι ε, με βάση και τις ανησυχίες που υπάρχουν ε, ε, θεωρούμε, για τη Γεωργία, θεωρούμε ότι πρέπει να, πιέσουμε, να πιέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Ρωσία να πληρεί τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στις συμφωνίες. Ε, πρέπει οι ε, θέσει τη ε, Ρωσία, των στρατιωτικών τη Ρωσία να παραμείνουν στα όρια που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο. Το ότι παραβιάζει την εντολή που έχει η Ρωσία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανισότητα, όπως είπα, στο πώς βλέπουμε εμεί τη λύση του προβλήματος και πώς τη βλέπουν οι υπόλοιποι. Η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Αποστολής ε, σε όλες τις περιοχές ε, θα δείξει ότι η Ρωσία ε, τηρεί τις συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ να σας απαντήσω και σε ερωτήματα αν υπάρχουν. Θα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λίζεκ. θα ήθελα να συζητήσω, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας για τις συζητήσεις στη Γενέβη. Είναι το μοναδικό μέρος στον οποίο ο διάλογος παραμένει εφικτός. Σας ευχαριστούμε για τις εκτιμήσεις που δώσατε για την κατάσταση. και να μας μιλήσετε σε λίγο για τη νέα στρατηγική την οποία θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνησή σας στα κατεχόμενα εδάφη. Νομίζω ότι ο πρόεδρος μας έθεσε τις ερωτήσεις τις οποίες θα ήθελα να θέσω, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα θέμα το οποίο ε, μπορεί να συζητηθεί εκ νέου. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας για τις πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε και για ένα σενάριο το οποίο μας περιέγραψε, το οποίο είναι σχετικά θετικό. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω Στην περίπτωση κατά την οποία το θετικό σενάριο πράγματι πραγματοθεί, πράγματι ολοκληρωθεί, πώς θα αντιδράσουν οι γεωργιανές αρχές. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι γεωργιανές αρχές τα κατεχόμενα εδάφη και αναφέρομαι σε επίπεδο πολιτικό βέβαια, όχι στρατιωτικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι και πριν τον πόλεμο υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στις τοπικές αρχές και σε κάποιες πολιτικές ομάδες στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Προβλήματα υπήρχαν και πριν από τον πόλεμο λοιπόν. Υπήρχαν συγκεκριμένες ομάδες, πολιτικές ή εθνοτικές, που είχαν συγκεκριμένες επιθυμίες για αυτονομία, για ανεξαρτησία, για απελευθέρωση εισαγωγικά από την γεωργία κτλ. Τώρα, τα σενάρια αυτοί, ε, τι ίχνη έχουν αφήσει στην πολιτική σκέψη στο Τμπιλίσι. Είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε ακόμα. Έχετε προβλέψει κάποιες πιθανές συνταγματικές ρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν μια βιώσιμη αυτονομία των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ. Μια στιγμή θα ακούσουμε τρεις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσετε ομαδικά. Η κυρία Κοπά. Thank you, President. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσκεκλημένο μας για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Οι συνέπειες του πολέμου είναι κάτι το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στη Γεωργία και κατανοούμε και υποστηρίζουμε την προσπάθεια της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η μοναδική αποστολή αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει επί πολύ την κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του έχει καταδικάσει τις ρωσικές επιθέσεις αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η βασική ευθύνη πέφτει και στις δύο πλευρές γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι υπήρξαν ατυχείς ενέργειες από τον πρόεδρο Σακασβίλη πριν από τη ρωσική επίθεση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο νομιμοποιεί τη ρωσική αντίδραση. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα γεγονότα και δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη μία πλευρά. Το θέμα είναι ποιες είναι οι προοπτικές της α, ε, ε, Γεωργίας σχετικά με τη μελλοντική υποψηφιότητά της. Πιστεύετε ότι η προοπτική αυτή υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες. Ξέρετε ότι γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σε αυτή τη φάση για τη νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ. Ε, πώς βλέπετε αυτή την δυνατότητα. Πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου θα τεθεί και το θέμα της υποψηφιότητας της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριο Λαντσμπέργης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά κάτι το οποίο είχε γίνει πριν δύο χρόνια. Είχαν δημόσια δηλώσει οι Ρώσοι ότι θα προχωρήσουν στην επέκταση ε, του ομοσπονδιακού εδάφους μετά από διμερή συμφωνία με το Συμβάλλη. έτσι ώστε να δημιουργήσουν περαιτέρω ε, ε, χώρους για εγκατάσταση εξοπλισμών για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς του Σότσι. Δεύτερη ερώτηση. Πώς αντιμετωπίζεται η Ρωσία στην συνάντηση της Γενέβης, σαν στρατιωτικός εισβολέας, Merci. Thank you, Chair. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε πάει στη Γεωργία πριν λίγες εβδομάδες για παρακολούθηση των τοπικών εκλογών. Και είχαμε τη δυνατότητα να πάμε και στον Γκόρι. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα των προσφύγων. και είναι απίθανο να μπορέσει κανείς να επιστρέψει στα εδάφη που κατέχει ως αιτία. Το 2008 πριν από τον πόλεμο γιατί η Γεωργία δεν επικαλέστηκε το άρθρο 4 της συνθήκης της Washington για συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την Επιτροπή ΝΑΤΟ Γεωργίας. Το Δεκέμβριο του 2008 οι Υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα ετήσιο πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Επιτροπής αυτής. Τι γίνεται ακριβώς με αυτό το πρόγραμμα, έχει προχωρήσει. Ε, ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω με τη σειρά. Πρώτον, η διαδικασία της Γενέβης. Παραμένει μοναδική δυνατότητα προσπάθειας έβρεσης πολιτικής λύσης. είναι το μοναδικό φόρουμ όπου έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και ελπίζω να προκαλεί και το ενδιαφέρον των άλλων. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια η οποία έχει ήδη γίνει είναι σημαντική. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι τα απτά αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε όλοι. Αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν τις συναντήσεις αυτές σημαντικές. Σε ευχαριστούμε για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και για τις προσωπικές παρεμβάσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρεμποδίσει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και απομακρύνει από τις πιθανές λύσεις. Όταν ξεκίνησαν συζητήσεις για συγκεκριμένα έγγραφα, όπως τα θέματα του εγγράφου που αφορούν την τοπική ασφάλεια, ε, εκεί η ρωσική αντίδραση ήταν παραπλανητική. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες αυτές πλήρως. Η ερώτηση σχετικά με το λεγόμενο θετικό σενάριο και τι πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε στο μέλλον. Ας προσπαθήσουμε να πάμε λίγο πίσω στα γεγονότα του 2008 και ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτά τα οποία έχει κάνει από τότε η Γεωργία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πριν τον πόλεμο και την εισβολή, είχαμε προτείνει ορισμένες λύσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Είχαμε προτείνει ένα ειρηνευτικό σχέδιο είχε υπάρξει γερμανική διαμεσολάβηση και γερμανική προσπάθεια και ο Υπουργός Εξωτερικών Στάινμαγερ είχε συνεισφέρει και αυτός, είχε ταξιδέψει στην περιοχή. Είχαμε προσπαθήσει να δείξουμε το τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε για να επιληθεί το πρόβλημα. Δυστυχώς απερίφθη η πρόταση αυτή γιατί το Κρεμλίνο δεν ήθελε εν πάση περιπτώσει μια τέτοια διαμεσολάβηση. Παρ' όλα αυτά διαμορφώσαμε μια σαφέστατη πρόταση και σχετικά με την συνταγματική επίλυση του θέματος, με την μέγιστη, ε, την ευρύτατη δυνατή μορφή αυτονομίας. ανάμεσα στη συγκεκριμένη περιοχή και το κέντρο και προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να έρθουμε σε επαφή, να πλησιάσουμε τις ενδιάμεσες αυτές αρχές στην Οσετία και στην Απχαζία. Υπήρξαν κάποιες απόπειρες διαπραγμάτευσης με το καθεστώς της Ρωσίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος είχε εμπλακεί σε αυτές τις προσπάθειες, αλλά δυστυχώς αυτός ο δρόμος δεν απέδωσε. Παρά τις δυσκολίες αυτές και παρά την εισβολή του 2008, συνεχίζουμε να προσπαθούμε να είμαστε θετικοί για τον ρόλο τον οποίο μπορούμε να αναλάβουμε και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση η οποία προβλέπεται στα πλαίσια της στρατηγικής της κυβέρνησης της Γεωργίας και τη σύνδεσή μας με τους πληθυσμούς των κατεχωμένων περιοχών. Η στρατηγική αυτή έχει γίνει δεκτή από τις υπόλοιπες δυνάμεις στη χώρα και έχει αξιολογηθεί θετικά και από φίλες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλες. Εγώ από εδώ θα πάω στο Παρίσι όπου θα έχουμε ε, πολύ σοβαρές συζητήσεις για το πρόγραμμα δράσης το οποίο συνοδεύει την στρατηγική στην οποία αναφέρθηκα. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένες επαφές έτσι ώστε να αποπολιτικοποιήσουμε την ίδια διαδικασία. Θέλουμε να προσφέρουμε συγκεκριμένα κίνητρα στον λαό της περιοχής, να φέρουμε σε επαφή τους κατοίκους της περιοχής σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και νομίζουμε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε θετικοί σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Αλλά από εμά εξαρτάται να είμαστε αποτελεσματικοί. γιατί όσο μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής που χωρίζεται από τη διαχωριστική γραμμή, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η λύση και τόσο περισσότερο θα εμβαθύνει η ρωσική παρουσία. Σχετικά με το τι προηγήθηκε της επίθεσης της εισβολής στη Γεωργία. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Μιλάμε για το ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο, το 2008. Πολλοί ξεχνούν να λέγουν, να πούν ε, τι ήταν πίσω από όλα αυτά. Κανένας δεν αναφέρθηκε στα διαβατήρια τα οποία είχαν διανύμει οι Ρώσοι. Κανένας δεν είχε μιλήσει για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία. Η ρωσική παρουσία ήταν εκεί μετά από παραβίαση της ειρηνευτικής διαδικασίας Κανένας δεν είχε μιλήσει για, την, για τους φόνους των γεωργιανών ειρηνευτών τον Νοέμβριο, στις 8 Νοεμβρίου του 2008. Κανένας δεν μιλάει για τα χωριά τα οποία βομβαρδίστηκαν από τις ρωσικές μονάδες, τις δίθεν ειρηνευτικές μονάδες, τις οποίες είχε προσφέρει σε εισαγωγικά η Ρωσία. Κανένας δεν είπε ότι η πολιτοφυλακή της Νότιας Οσετίας χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που τους είχαν δώσει οι Ρώσοι. Και όταν μιλάμε για την εκκίνηση του πολέμου θα πρέπει να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και εμείς δείξαμε πώς είχαν γίνει τα πράγματα, είχαμε δείξει πώς οι τακτικές ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κυρίαρχο έδαφος της Γεωργίας πριν ξεκινήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις. Κανένας δεν αναφέρεται γι' αυτό. Ακόμα και οι αξιωματούχοι της Ρωσίας ε, το παραδέχονται αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός έχουμε όλο και περισσότερες αποδείξεις από τους στρατιώτες οι οποίοι ήταν εκεί εγκατεστημένοι από τα γράμματα που έστελναν στους γονείς τους. Κανένας δεν μιλάει για τις στρατιωτικές ασκήσεις τις οποίες έκανε η Ρωσία πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, οι οποίες ε, προέβλεπαν το συγκεκριμένο σενάριο το οποίο εξελίχθηκε. Και αν κοιτάξει κανείς την συγκεκριμένη έκθεση από πλευράς Ρωσίας θα τα επιβεβαιώσει όλα αυτά. Η ίδια αυτή προπαγάνδα είχε διαταχθεί πριν από τον πόλεμο πώς είχαν μοιραστεί εγχειρίδια στους ε, Ρώσους της περιοχής, πώς ε, τους είχε ζητηθεί να προσπαθήσουν να, προκαλέσουν, να προκαλέσουν προκλήσεις στην περιοχή. Όταν λοιπόν βλέπει κανείς το ποιος ε, έριξε την πρώτη σφαίρα θα πρέπει να δει τι προηγήθηκε. Δεν μπορεί να αγνοήσει το τι προηγήθηκε. Αυτά τα λίγα για τα θέματα της γεωργίας. Και να πω και κάτι άλλο σχετικά με τον πόλεμο. Ε, πράγματι η Γεωργία δεν εισέβαλε καμία άλλη περιοχή. Ε, μιλάμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν σε κυρίαρχο γεωργιανό έδαφος. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να τα καταλάβει κανείς. Σχετικά με τις προσδοκίες μας και τις φιλοδοξίες μας σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με τον ΝΑΤΟ σε επίπεδο διμερές, το NGC το λεγόμενο. Έχουμε ένα πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τη Γεωργιανή κυβέρνηση και τις συμμαχικές δυνάμεις αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε έτσι ώστε να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας με τις απαιτήσει του ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε θετικά τα προβλήματα και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική της ανοιχτής φύρας από πλευράς του ΝΑΤΟ στη συνάντηση της Λισαβόνας το Νοέμβριο. η πολιτική αυτή είναι θετική. Έχουμε το παράδειγμα του Μαυροβουνίου και το παράδειγμα της Βοσνίας που το επιβεβαιούν. Αυτές είναι και οι πολιτικές φιλοδοξίες που έχουν οι Γεωργιανοί. Σχετικά τώρα με τις συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η Ρωσία, πράγματι έχουν συναφθεί τρεις συμφωνίες με τις τοπικές κυβερνήσεις, σε εισαγωγικά κυβερνήσεις, και σχετικά με την στρατιωτική τους παρουσία. Όπως γνωρίζετε, η Ρωσία μονομερός και κατά του διεθνούς δικαίου, αντίθετα με το διεθνές δίκαιο, έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των κατεχομένων αυτών περιοχών και έχει συνάψει συμφωνίες με τις περιοχές αυτές, όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά και σε επίπεδο οικονομικής συνεργασίας και σε σχέση με τις αερομεταφορές θέλουν να νομιμοποιήσουν τις αερομεταφορές μεταξύ των δύο περιοχών χωρών και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η δυσαρέσκεια παρόλα αυτά είναι πολύ μεγάλη. Αν πιστεύει κανείς ότι οι Αμπχάζοι είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουν προχωρήσει οι εξελίξεις, κάνουν λάθος οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν ότι χρησιμοποιείται η περίπτωσή τους από την υπερδύναμη προς το δικό της υφέρον και δημιουργείται μια κάποια δυστημία και αυτή η δυστημία θα συνεχιστεί στο μέλλον. σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευρά μας της Ρωσίας σαν στρατιωτικού εισβολέα. Προφανώς η απόφαση τολμηρή την οποία υιοθέτησε το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας και το ευχαριστούμε γι' αυτό, δίδει μια νομική διάσταση θα έλεγα στην εισβολή της Ρωσίας στις χώρες της Δύσης έτσι ώστε να ονοματίζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που πρέπει. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα υπόδειγμα του τι μπορεί να ονομαστεί επίθεση και εισβολή στον 21ο αιώνα εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την κατάσταση η οποία υπάρχει και γι' αυτό ευχαριστώ τους Λιθουανούς φίλους. Τώρα, τα στρατόπεδα IDP. Ξέρουμε ότι δεν είναι για τους πρόσφυγες, δεν είναι η καλύτερη λύση. Η γεωργιανή κυβέρνηση έχει προσπαθήσει με τον ταχύτερο τρόπο να καλύψει τις ανάγκες και να προστατεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Οι συνθήκες είναι απλά ανεκτές. και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για να καλύψουμε τις οικιστικές τους ανάγκες. Δεν θα το είχαμε πετύχει αυτό χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια η οποία μας δόθηκε, αλλά και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Προσπαθούμε να σταθούμε απέναντι στα προβλήματα αυτά θετικά έτσι ώστε τα πράγματα να επανέλθουν σε ένα κανονικό ρυθμό. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κάποια δυστημία στον πληθυσμό αυτό, υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα όπως ανεργία, αλλά εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τα NGC. Τα NGC είναι η βασική μορφή συνεργασίας ανάμεσα στη Γεωργία και τον ΝΑΤΟ. και θα προσπαθήσουμε τον μηχανισμό αυτό να τον εξορθολογήσουμε ακόμα περισσότερο. Βοηθά τον ΝΑΤΟ σε κάποιους τομείς όπως σαν παράδειγμα την αναθεώρηση της, ε, τον έλεγχο μάλλον της κατάστασης στον τομέα της τάξης και ασφάλειας στη Γεωργία. Μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει πολλά απτά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε αποτελέσματα τέτοιου είδους. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε ένα τελευταίο ερώτημα του κ. Μπουτικόφου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ποκίτσε, ε, θεωρώ ότι είμαι φίλος της Γεωργίας αλλά ορισμένα από τα θέματα αυτά με, μου δημιουργούν απορία. Είπατε να τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα. Λοιπόν, αν έχετε συνέπεια με αυτό θα πρέπει να έχετε το θάρρος να πείτε ότι εμείς ξεκινήσαμε να πυροδοτούμε και όπως είπε κάποιος ε, γνωστός ε, ε, Γάλλος δεν ήταν κάτι παραπάνω από έγκλημα, ήταν ένα κουτό λάθος. Γιατί λοιπόν δεν σέβεστε το γεγονός τα μέλη αυτού του κοινοβουλίου, για παράδειγμα, είπαν, αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα στα οποία εμπενιχθήκατε. Είπατε κανεί δεν μιλάει για τα διαβατήρια. Τουλάχιστον αυτό δεν είναι αλήθεια για το κοινοβούλιο μας. Κανεί δεν μιλάει για αυτό, για αυτό και τούτο και τ' άλλο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν νομίζω ότι βοηθάτε την υπόθεσή σας ε, τα άτομα με τον τρόπο που κάνετε τα πράγματα. Δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Εσείς είσαστε άσπροι και το Κρεμλίνο είναι μαύρο. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, πιο περίπλοκα. Και ε, ορισμένα από τα όσα λένε ε, ε, οι Γεωργιανοί περιπλέκουν τα πράγματα. Η μια εσωτερική ανάλυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μας λέει ότι θεωρεί ότι η πολιτική ρητορική από κάθε πλευρά είναι προκλητική τι προτείνετε λοιπόν εσείς για να αλλάξει αυτή η κατάσταση από πλευράς Γεωργίας. Και δεύτερο ερώτημα. Συμφωνείτε με την ανάλυση του Συμβουλίου ότι η επανέναρξη των ενόπλων εχθροπραξιών είναι απίθανη μεν, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο. Ευχαριστώ, πρέπει να ολοκληρώσουμε, η Αντιπρόεδρος. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει σχέση με την αλλαγή του συντάγματος. Ξέρω ότι μόλις τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Σχεδιάζεται να, ε, να κάνετε κάτι σε σχέση με την Απχασία και την Αθιοσετία. δηλαδή τι προβλέπετε μια, ε, ε, ένα τύπο ομοσπονδίας, Επίσης έχετε την δημόσια υποστήριξη για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Ε, προβλέπετε κάτι σχετικό σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Φοβούμαι ειλικρινά ότι θα γίνεται η επόμενη Κύπρος. Thank you, Chairman. Ε, Απλά θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο περισσότερα σχετικά με ε, την, την εμπλοκή σε αυτά τα εδάφη. Ε, ε συναντήσαμε νέους εκπροσώπους ε, και από τη Γεωργία και από την Νότια Οσετία στα πλαίσια ενός προγράμματος των ΜΚΟ και φυσικά συζήτησαν. Δεν ήταν εύκολη συζήτηση, αλλά πώς σχεδιάσετε να δώσετε συνέχεια σε αυτή τη νέα στρατηγική επειδή παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή για να δούμε αν θα υπάρξει υλοποίηση, αν δεν θα παραμείνουν τα πράγματα ε, στα λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα και για ορισμένες συμβουλές που μας δώσατε. Νομίζω ότι δεν είπα ότι κανεί δεν δίνει προσοχή σε αυτά τα γεγονότα. Ξέρω ότι υπάρχουν σμένοι που αποδίδουν μεγάλη προσοχή στα γεγονότα. Τώρα, αν δούμε την ανατομία των εχθροπραξιών, η αναφορά που έκανε ήταν η εξή, ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα από ολιστική σκοπιά. Δεν λέω ότι κανένας ε, δεν έχει κάνει σφάλματα, αλλά πρέπει να δούμε το ιστορικό, να δούμε όλη την εικόνα γενικά. Πρώτα απ' όλα, οι εχθροπραξίες δεν ξεκίνησαν, όπως πιστεύετε, στις 8. Ε, οι ειρηνευτικές μονάδες της Γεωργίας σκοτώθηκαν στις 4 Αυγούστου και αυτό έγινε από ορισμένα στοιχεία τα οποία δεν ανήκαν στον τακτικό στρατό και υποστηρίχθηκαν από ορισμένε ρυθμίσεις. Αυτό υπάρχει εγγράφους. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Επίσης υπάρχουν τεκμήρια ότι, τα, ότι χωριά της Γεωργίας βομβαρδίστηκαν από μηχανισμούς που, εξοπλισμούς που δεν ήταν στη διάθεση των τοπικών εκπροσώπων. Και επίσης υπάρχουν τεκμήρια ότι αυτοί οι βομβαρδισμοί συνέβησαν από θέσεις που τότε ε, κατήχοντο από τους λεγόμενους ειρηνευτές των Ρώσων. Επίσης έχουμε ε, τεκμήρια για το πώς οι μονάδες, ε, οι μονάδες των Ρώσων συντόνιζαν τα πράγματα και γνώριζαν πού έπρεπε να γίνουν οι βομβαρδισμοί. Όλα αυτά είναι στοιχειοθετημένα. Και αυτό είναι γεγονός. αν θέλετε, έχουμε τα στοιχεία στη διάθεση μεταξύ σας. Ε, δεν πρέπει να έχετε την εντύπωση ότι δεν είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη που μας δίνετε. Είμαστε ευγνώμονες ε, και άλλωστε αυτό το ανέφερα και θα έχουμε πάντοτε αυτό το πνεύμα. Τώρα για το νέο σύνταγμα. Το νέο σύνταγμα ε, είναι σε μια διαδικασία που ξεκίνησε πέρσι και περιλαμβάνει έναν τομέα πολιτικών δυνάμεων, δεν περιλαμβάνει τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και η Επιτροπή συντονίζει τις προσπάθειες με τις χώρες εταίρους και εκείνες που ενδιαφέρονται ε, για να δώσουν το παρόν στη Γεωργία. Σε αυτή τη διαδικασία δεν συμμετέχει η κυβέρνηση. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Δεν είναι ο κλάδος μου δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται συζήτηση, είναι μια διαδικασία που συζητείτε και είμαι βεβαίως ότι θα δημοσιοποιηθεί, θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα. Αλλά η ίδια διαδικασία έχει αρκετή διαφάνεια για να εκπροσωπεί διαφορετικές απόψεις. Τώρα για τη δημόσια υποστήριξη στην προσχώρηση του ΝΑΤΟ θα έλεγα το εξής. Το 2008 η δημόσια υποστήριξη για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ ήταν μεγάλη. Νομίζω 70, 72, 74, πολύ μεγάλη αποδοχή και αυτή η τάση διατηρείται θα έλεγα. Και υπάρχει λοιπόν δημόσια υποστήριξη για προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Τι γίνεται για να διατηρηθεί. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα κέντρο ενημέρωση για θέματα ΝΑΤΟ ε, και υπάρχει μια εκστατεία ευαισθητοποίηση του κοινού και υπάρχει υποστήριξη για την διαποδαγώγηση του κοινού, για την ενημέρωση του κοινού, για τα πλεονεκτήματα ε, που θα προκύψουν από την προσχώρηση στον ΝΑΤΟ. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ναι, υπάρχει ενημέρωση και υποστήριξη από το κοινό. Τώρα, το ερώτημα σχετικά με την στρατηγική την που την οποία έχουμε προτείνει συμφωνώ ότι δεν πρέπει να είναι μόνο δημόσιες σχέσεις και λόγια. Πρέπει να γίνει κάτι στην πράξη. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε η στρατηγική. Το πρώτο που κάναμε ήταν ότι ενημερώσαμε σχετικά την κοινωνία των πολιτών και τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Συνεπώς είδαμε ποια ήταν η αντίδρασή τους και Όλα αυτά τα σχόλια περιλήφθησαν στη στρατηγική. Κατόπιν προχωρήσαμε σε ένα άλλο στάδιο. Συζητήσαμε τη στρατηγική με τους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας στη Γεωργία μέσω των ε, πρεσβειών ε, για να ενημερωθούν και οι κυβερνήσεις, αλλά και με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε ένας ειδικό εκπρόσωπος και επίσης ορισμένοι γνωστοί εμπειρογνώμονες από τη Γερμανία, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και τελικά η στρατηγική στέφθηκε με επιτυχία επειδή δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, αν θέλετε, για όλους, ώστε να σκέφτονται θετικά το επόμενο βήμα. Τώρα, για το σχέδιο δράσης, που είναι κάτι το πιο συγκεκριμένο, όχι μόνον Μιλάμε για τις δημόσιες σχέσεις, ε, δεν μιλάμε μόνο, δεν είναι μόνο λόγια, αλλά φτάσαμε σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την υλοποίηση της στρατηγικής. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, τι συνεπάγεται. Θα σας δώσω τι λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να σας δώσω και το ίδιο το σχέδιο δράσης Όπω σα είπα, θα μεταβώ στο Παρίσι, μετά από εδώ θα έχουμε μια συνάντηση με τι κυβερνήσει εταίρου αλλά και τι σχετικέ οργανώσει. Θα συζητήσουμε το θέμα και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο δράση. Το σχέδιο δράση αναφέρεται στη δημιουργία ε, ε, ε, κινήτρων ώστε να συμμετάσχει ο πληθυσμό, Μιλάμε για ένα κοινό οικονομικό χώρο, να δημιουργηθεί μια αγορά όπου θα μπορεί κανεί να πουλάει αγαθά, να γίνονται αγοραπολισίε αγαθών. Επίσης, πρέπει να σας πούμε ότι οι τιμές στην Απχαζία είναι πολύ ψηλές. Πώς να σας το πω. Είναι ένα κράτος με διαφθορά που δίκεται από μια ελίτ με παράδοξες σχέσεις μεταξύ του. Το κόστος μεταφοράς είναι πολύ ψηλό. Γι' αυτό θέλει ο κόσμος πραγματικά να κάνει κάτι. Τώρα, άλλα. Θα προσφέρουμε μια, ε, κοινωνικές υποδομές. υγεία, για παράδειγμα. Όπως σα είπα, οι τιμέ είναι πολύ υψηλέ και το σύστημα υγείας ε, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ε, πολλοί, πολλοί πηγαίνουν στη Γεωργία από την Απτυχαζία. Πολλοί. Ε, θα υπάρξει μια γενική συζήτηση, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως θα τίνουμε χείρα κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τις εξηγήσεις που δώσατε και για το γεγονός ότι απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μας για τη Γεωργία στα πλαίσια της αποστολής UMM. Ça marche. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μα τώρα. Θα ήθελα να χαιρετήσω μία αντιπροσωπή αξιωματούχων από την Bundeswehr. Επίσης θα ήθελα να σα διευκρινίσω για όσους έχουν ερωτήματα ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία σύντομα ελπίζω, να έχουμε μια συζήτηση με Ρώσους εκπροσώπους, όχι μόνο για το θέμα της Γεωργίας φυσικά, μας χρειάζεται ένας διάλογος ευρύτερος ε, και θα συναντήσω τον πρέσβη κ. Τσίζοφ και ελπίζω ότι θα έχουμε την ε, ευκαιρία να οργανώσουμε μια συνάντηση στα πλαίσια της υποπιτροπής ώστε μεταξύ των άλλων να μιλήσουμε για το θέμα της γεωργίας αλλά και για πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Καλωσορίζω λοιπόν τον, τον πρέσβη κ. Χάμπερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, αποστολής παρακολούθησης στη Γεωργία και ο κ. Χάμπερ έρχεται συχνά εδώ εφόσον εξετάζουμε τις διάφορες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν θέλω να κάνω μια ιστορική υπόμνηση για τις ε, συνθήκες ανάπτυξης ε, της αποστολής της UMM στη Γεωργία. Απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μετά από την απόσταση του ΩΣΑ των Ηνωμένων Εθνών, η αποστολή παρακολούθησε η UNM είναι η μόνη διεθνή παρουσία στη Γεωργία που παρακολουθεί τα πράγματα και τα πράγματα που διαμορφώθηκαν μετά από τα γεγονότα του Αυγούστου 2008. Αυτή η αποστολή είναι πολύ σημαντική, περιλαμβάνει πάνω από 250 άτομα και ελπίζω ότι θα διατηρηθεί αυτό το επίπεδο. Επ' αυτού θα ήθελα να ε, χαιρετήσω το γεγονός ότι παρατάθηκε για ένα χρόνο ε, η αποστολή αυτή έχει σχεδόν αποφασιστεί επισήμω, αλλά λογικά θα αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή δύσκολη φυσικά, είναι μια αποστολή που αντιμετωπίζει δυσκολίες επί τόπου και δυστυχώς μη σεβασμό ε, όλων των πλευρών της αποστολής από ορισμένους. Ζείτε λοιπόν σε ένα περιβάλλον ευαίσθητο, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με την αποστολή σας, με την εντολή σας και το τι περιμένουμε. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Καμπανάουρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να περάσω στα, να περάσω στα αγγλικά. Κυρίε και κύριοι, να σας πω κάποια πράγματα για, για μια από τι πιο επιτυχημένε αποστολές. Πρέπει να πω ότι θέλουμε να υπάρξει σταθεροποίηση στην Γεωργία και να λυθούν επιτέλους αυτές οι διενέξει που υπάρχουν. Η αποστολή, η πολιτική, είναι η πιο απτή απόδειξη της δέσμευσης που δείχνουμε. Όπως ξέρετε, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις πιο ορατές, από τις πιο επιτυχείς ε, αποστολές και μετά από, την, ε, από τη συμφωνία το 2008 για την, ε, με, μεταξύ Σαρκοζή και Μετβέντεφ ε, εφαρμόζεται που, με τρόπο τέτοιο που πολλές φορές ε, ε, προσπαθεί να ξεπεράσει τα, τα εσκαμένα. Ο πρέσβης ε, Χάρμπορ θα σας αναφέρει κάποια πράγματα για την αποστολή και πώς ο ίδιος βλέπει τα πράγματα εκεί επί τόπου. Σε στρατηγικό επίπεδο να υπενθυμίσω ότι η Ρωσία ακόμη δεν συμμορφώνεται με το σχέδιο έξι σημείων που, ζητά να αποσύρει τις, ε, τις στρατιωτικές δυνάμεις ε, στις, στα όρια που είχαν πριν από, την, από το βόλεμο. Και βεβαίως σε κάποια σημεία διέλευσης ιδιαίτερα χρειάζονται τη δική μας προσοχή. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλους τους ε, συνομιλητές μας ε, και τους εταίρους μας, ελπίζοντας να μπορέσουμε να πιέσουμε ε, τη Ρωσία να αποσυρθεί. Ελπίζουμε να το κάνετε και εσείς. Παρά την επιτυχία της, η αποστολή είναι συγκεκριμένα πράγματα αυτά που μπορεί να κάνει. Η πολιτική πρόοδος προς μια πολιτική επίλυση της διένεξης είναι η μόνη δυνατότητα για να υπάρξει σταθερότητα. Η πρόοδος, παρόλο που είναι περιορισμένη στην Γενέβη, υπάρχει και επιμένουμε ότι η διαδικασία της Γενέβης να παραμείνει το μοναδικό φόρουμ όπου εκπροσωπούνται όλα τα μέλη. Θεωρούμε ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική για την περιοχή και όπως είπα και ο πρόεδρος μόλις, ε, περιμένουμε ολοκλήρωση της πολιτικής συμφωνίας για την επέκταση της, απο... της αποστολής μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011. Και τώρα να δώσω το λόγο στον, στον πρέσβη Χάρμπορ και να πω ότι προσβλέπουμε στην δική σας συμβολή στην ε, περιοχή. Πριν δώσω το λόγο στον Χάμπερ, πράγματι μια αντιπροσωπεία της ε, υποεπιτροπής μας θα πάει πολύ σύντομα στη Γεωργία και ο κύριος Λίζεκ θα πάει και αυτό στη Γεωργία, αντιπρόεδρος, είναι εισηγητής για τη Γεωργία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που μπορώ να σας ενημερώσω για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποστολή αυτή. Προσβλέπουμε στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας σας τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη υποδεχθεί κάποιους από εσά πέρυσι. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη και το ίδιο θα ισχύσει και για την επόμενη. Οι περισσότεροι επισκέπτες στην περιοχή είναι ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν επί τόπου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα πράγματα σύμφωνα με την εντολή μας. Πρώτον, σταθεροποίηση, εξομάλυνση, μέτρα εμπιστοσύνης και ε, συνεισφορά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το τελευταίο κομμάτι δεν είναι κάτι το οποίο θα θίξω εγώ. Εμείς ενημερώνουμε όσο μπορούμε και είναι σχετικά ικανοποιημένοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μας. Πρώτον, σταθεροποίηση. Σταθεροποίηση είναι η βασική μας επιτυχία από την αρχή της αποστολής αυτής. Η κατάσταση στα πλαίσια των, των διοικητικών συνόρων Τη διοικητική συνοριακή γραμμή καλύτερα γιατί δεν είναι διεθνώ αναγνωρισμένα τα σύνορα, βελτιώνεται συνεχώ Όταν φτάσαμε στο θέατρο των επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο του 2008 και αναλάβαμε τις περιπολίες στις αρχές του 2009 και οι Γεωργιανοί και οι Ρώσοι, συνομιλητές μας εκείνη την περίοδο, αναφέρθηκαν στις προσδοκίες τις οποίες είχαν ε, ότι έπρεπε σε λίγες εβδομάδες να αρχίσουν εκ νέου οι εχθροπραξίες. Οι Γεωργιανοί πίστευαν ότι οι Ρώσοι δεν τέλειωσαν τη δουλειά τους, οι Ρώσοι πίστευαν ότι οι Γεωργιανοί δεν ήταν ικανοποιημένοι από την κατάσταση και θα προσπαθούσαν να την αλλάξουν βία. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Υπήρξαν συγκεκριμένα επεισόδια κατά, τη, κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής και κυρίως υπήρξαν επιθέσεις στις βάρος γεωργιανών αστυνομικών. Όταν φτάσαμε εκεί στις 12 Αυγούστου, είχαν σκοτωθεί έξι γεωργιανοί αστυνομικοί, μετά την άφηξή μας ε, φωνεύτησαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 και από τότε δεν έχουμε ε, απώλειες σε επίπεδο μη μάχημου πληθυσμού. Αυτή είναι η κατάσταση της έκφρασης βίας κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής, της διοικητικής αυτής διαχωριστικής γραμμής. Υπάρχει σαφέστατη μείωση της έντασης, δηλαδή μετά την ανάπτυξη των δυνάμεών μας. Έχουμε κάποια μέσα για την εφαρμογή της σταθεροποίησης. Καταρχάς υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης που υπογράψαμε με το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας. Με το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τη στιγμή αναλάβαμε περιπολίες. Ήταν μαζί μας ο Κλόκμα και συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Γεωργίας τον τρόπο που θα κάναμε τη δουλειά μας. Αυτό το μνημόνιο κατανόησης, αμοιβαίας κατανόησης αφορά τη στελέχωση των αστυνομικών φυλακίων. Οι Γεωργιανοί υποχρεούνται να μας ενημερώνουν για τις ενέργειές τους, να υπάρχει διαφάνεια από πλευράς τους και υπάρχει και μία θερμή γραμμή θα έλεγα ή μάλλον όχι, θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Μετά από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες παρετάθησαν μετά τον Ιανουάριο του 2009 υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας και στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας αποκτήσαμε το δικαίωμα επιθεώρησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα στην περιοχή η οποία συνορεύει άμεσα στην διοικητική διαχωριστική γραμμή ο πιο σημαντικός βασικός τομέας είναι στην περιοχή της κοιλάδας του Αραγκούρε, πολύ κοντά στον Τμπιλίσι, 50 χιλιόμετρα από τον Τμπιλίσι. Υπάρχει ένα μεγάλο ρωσικό στρατόπεδο και εκεί υπάρχει η δυνατότητα κάποια στιγμή πολύ εύκολα να ξεκινήσουν θα έλεγα εχθροπραξίες. Προσπαθούμε λοιπόν να περιορίσουμε εμείς τη συγκέντρωση βαρέως εξοπλισμού και στρατευμάτων στην περιοχή αυτή της ε, Αμπχαζίας και της Νότιας ε, Οσετίας. Και αυτό πέραν των υποχρεώσεων τις οποίες έχουν αναλάβει στα πλαίσια της Συμφωνίας των Έξι Σημείων. Οι προσπάθειές μας στέφθηκαν από επιτυχία. Τους μήνες μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου, είχαμε κατηγορηθεί από πλευράς των Ρώσων και από πλευράς της Νότιας Οσετίας ότι υπήρξαν κατηγορίες ότι οι Γεωργιανοί μάζευαν στρατεύματα έτσι ώστε να επιτεθούν και να έρθουν σε σύγκρουση με αυτούς. Εμείς τα διαψεύσαμε, τα ελέγξαμε και τα διαψεύσαμε και κάποια στιγμή σταμάτησαν όλες αυτές, όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί και από τότε δεν έχουν ξαναγίνει, από το καλοκαίρι του 2009. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν για τη σταθεροποίηση της κατάστασης. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δική μας παρουσία, αλλά φυσικά και οι εμπλεκόμενοι στη σύραξη θέλουν τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν. Η συνεργασία μας με τις γεωργιανές αστυνομικές δυνάμεις και με το Υπουργείο Άμυνας είναι καλή, οφείλεται στο ότι επίσης στην παρουσία των Ρώσων συνοριοφυλάκων. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμά τους να είναι εκεί βέβαια, γιατί βρίσκονται εκεί ανάμεσα, εκεί μετά από συμφωνία που υπέγραψε η τοπική συσσαγωγικά κυβέρνηση με τους Ρώσους αλλά παρόλα αυτά αποτελεί ένα σημείο βελτίωσης σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση όπου είχαμε να κάνουμε με ατάκτους πολύ συχνά μεθυσμένους, ανεξέλεγκτους οι οποίοι ε, περιπολούσαν κατά μήκο της διαχωριστικής διοικητικής γραμμής. Λοιπόν, με τους Ρώσους συνοριοφύλακες η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Το 1 τρίτο των παρατηρητών μας λοιπόν εμπλέκονται στην προσπάθεια σταθεροποίησης κατά μήκος της γραμμής αυτής. Νομίζω ότι η βασική προσφορά μας η βασική συνεισφορά μας, συγγνώμη, and seen Έχουμε βοηθήσει να υπάρξει ένας διαχωρισμός στις επαφές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ε, ε, επεισόδια. Η κατάσταση είναι σχετικά ήρεμη, αλλά δεν έχουμε εγγυήσει για την παραμονή αυτής της ηρεμίας και είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η γεωργιανή κυβέρνηση δείχνει να εκτιμά την προσπάθειά μας. Μας λέγει επίσημα ότι χωρίς την παρουσία μας η κατάσταση και η σταθερότητα στην περιοχή γύρω από την διαχωριστική γραμμή θα ήταν πολύ χειρότερη. Στρέφοντας το βλέμμα προς τα πίσω λίγο, μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε και πιο πριν, Νομίζω ότι διαψέστησαν οι ισχυρισμοί αυτών που το 2009 έλεγαν ότι θα εντατικοποιηθούν οι εντάσεις ακόμα περισσότερο και θα έχουμε νέες σειράξεις κτλ. Νομίζω ότι η αξία της αποστολής μας επιβεβαιούται από, τη διάψευση αυτών των ισχυρισμών. Τώρα, η εξομάλυνση της κατάστασης είναι η δεύτερη μας αποστολή. Ε, ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ σαφές εξ αρχής. Έπρεπε να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε με κάποιο τρόπο. Όπως γνωρίζετε, ο πόλεμος οδήγησε σε μετακίνηση 100.000 ανθρώπων περίπου στη νότια Οσετία γύρω από την πόλη Γκόρη. Κάποιοι επέστρεψαν στην περιοχή τους, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετές χιλιάδες που δεν είχαν μπορέσει να επιστρέψουν, ιδιαίτερα μετά από ε, τον έλεγχο τον ρωσικό όταν ανέλαβαν οι Ρώσοι να ελέγχουν τη λεγόμενη ενδιάμεση ζώνη. Ε, έγινε προσπάθεια όμως ε, ενίσχυσης της επιστροφής αυτής και νομίζω ότι ουσιαστικά κάναμε κάποια πρώτα θετικά βήματα. Υπάρχουν βέβαια αρκετές δεκάδες χιλιάδες ακόμα ανθρώπων που από την Νότια αιτία δεν μπορούν να επιστρέψουν με εξαίρεση τους κατοίκους της κοιλάδας του Αραγκούρη, όπου εκεί η ελευθερία επανεγκατάστασης είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι στις υπόλοιπες περιοχές. Όπως γνωρίζετε, δεν υπήρξαν ε, πρόσφυγες από την Αμπχαζία εκτός ε, από την περιοχή του Αχαγκούρη. Έγινε σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούσαν να επιστρέψουν και η γεωργιανή κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα σε μεγάλη κλίμακα για να τους εγκαταστήσει και να τους ενσωματώσει στην ε, ε, γεωργιανή κοινωνία. Μεταφέραμε λοιπόν εμείς την παρατήρησή μας από την αποστολή εξομάλυνσης στην αποστολή παρατήρησης αυτού του πληθυσμού Προσπαθήσαμε να δούμε πώς πηγαίνει η κατάσταση για την επανεγκατάστασή τους και ε, ενημερώνουμε συστηματικά για τις εξελίξεις την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία χρηματοδοτεί τα προγράμματα των προσφύγων αυτών. Υπάρχουν πρόσφυγες και από τις πολεμικές συγκρούσεις της δεκαετίας του 90 κυρίως από την Αμπχαζία και όχι τόσο από την Νότια Ουσετία. Εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα προσφύγων και ε, ελέγχουμε την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος και σε αυτούς. Το 1 τρίτο των παρατηρητών μας ασχολείται λοιπόν με τα θέματα των προσφύγων. Βέβαια η υπόθεση αυτή έχει αρχίσει ε, να βρίσκεται σε μια κάποια στασιμότητα θα έλεγα. Επισκεπτόμεθα τις περιοχές εγκατάστασης ε, και τα στρατόπεδα των προσφύγων, ζητάμε από τον κόσμο να μας πει τις απόψεις τους, μας έχουν γνωρίσει αρκετά, δεν, τα πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτή τη φάση για τους πρόσφυγες και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα μεταξύ των οποίων να διασφαλίσουμε και την ελευθερία διακίνησης πέραν της γραμμής της διαχωριστικής. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω για τη γεωργιανή στρατηγική για τα κατεχόμενα εδάφη. Ενημερωθήκατε από τον κύριο Φωστίτσε γι' αυτό είναι μια πολιτική, θα έλεγα, η οποία στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πολιτικό έγγραφο, αν δει την ιστορία της σύγκρουση, και έχει νομίζω την δυνατότητα να βελτιώσει την κατάσταση και να εξομαλύνει τα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι ενημερωθήκατε λεπτομερώς. Η ελευθερία διακίνηση και ελεύθερη κυκλοφορία στην περιοχή της συνοριακής αυτής διοικητικής γραμμής είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις γεωργικές δραστηριότητες και έχουμε αρκετές ιδέες έτσι ώστε η, γραμμή αυτή να γίνει πλέον πορόδης ε, για τους ε, άμπαχους πληθυσμούς. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις της γεωργιανής στρατηγικής, οι οποίες ε, δεν προϋποθέτουν επιπλέον κόστος, απλά προϋποθέτουν κάποιες διοικητικές αλλαγές, σχετικά με την αναδιάταξη των αστυνομικών δυνάμεων της Γεωργίας. Είμαστε σε στενή επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών και έχουμε διάλογο μαζί τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πολλές και διαφορετικές ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί την τάξη και την ασφάλεια διαφορετικές από τις δικές μας. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει πρόοδος και εκεί. Και τέλος υπάρχουν τα θέματα οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η οικοδόμηση των μέτρων εμπιστοσύνης γιατί η σταθεροποίηση από μόνο της απλά θα παγώσει τη σύγκρουση. Οι εμπειρίες μας από το 90 δείχνει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Ε, μια τέτοια παγωμένη σύγκρουση θα ξεσπάσει ξανά. Ξέρουμε επίσης ε, και την εμπειρία που έχει ο ΩΣΑ ο ΑΣΕ μάλλον, συγγνώμη, ο ΑΣΕ στην περιοχή και πίστευαν ότι έλεγχαν την κατάσταση παρόλες τις παρεμβάσεις τους, αλλά τελικά η κατάσταση ξέσπασε με τραγικές συνέπειες τον Αύγουστο του 2009. Αν δεν καταφέρει κανείς να αντιμετωπίσει τις υποβόσκουσες αιτίε μιας τέτοιας σύγκρουσης, προφανώς η σταθεροποίηση από μόνη της δεν βοηθάει πάρα πολύ. Η οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνη. Αρχίσαμε να τα αντιμετωπίζουμε σαν θέματα μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις επαφές ανάμεσα σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τις δύο πλευρές. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε και εξακολουθούμε να μην έχουμε πρόσβαση στην άλλη πλευρά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία των πολιτών είναι αρκετά ασθενής στη Γεωργία και ακόμα πιο ασθενής στην Νότια Οσετία. Ίσως τα πράγματα να είναι λίγο διαφορετικά στην Απχαζία. Αλλά για την περιοχή Γκόρη υπάρχει πρόβλημα. Γιατί εκεί κατοικούν εθνοτικά Γεωργιανοί στην πλειοψηφία τους. Δεν έχουμε λοιπόν ισχυρού, δεν είχαμε ισχυρού εταίρους με τους οποίους να συνομιλήσουμε. Αλλά ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει τη Γενέβη και δημιούργησαν τον λεγόμενο μηχανισμό πρόληψης και ανταπόδοσης. Υπάρχουν δεκαπενθήμερες λοιπόν συναντήσει, προβλέπονται στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού στην Απχαζία υπό, τις των υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην Απχαζία των ε, κατοίκων της περιοχής, των Ρώσων, των Γεωργιανών και συζητάμε θέματα που δημιουργούνται στον τομέα της ασφάλειας για να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα. Οι Απχάζοι πήραν πολύ χρόνο για να φτάσουν σε αυτό το μηχανισμό, αλλά κάθε δύο-τρεις εβδομάδες συναντώμεθα, η ατμόσφαιρα βελτιώνεται συνεχώς, υπάρχουν εμπιστευτικές συνομιλίες στα περιθώρια των συναντήσεων αυτών, και αυτό είναι κάτι το γενικότερα θετικό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όμως ότι η αντιμετώπιση του θέματος ασφαλείας και από τις δύο πλευρές είναι μονομερής. Θέλουν να διασφαλίσουν την ασφάλεια στην περιοχή η οποία φτάνει μέχρι τη διοικητική γραμμή και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια λήψης μέτρων συλλογικής ασφάλειας και από τις δύο πλευρές. Εμείς προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε τους τομείς, τους τομείς τους οποίους θα υπάρξει δυνατότητα συνεργασίας, αλλά δεν το έχουμε πετύχει, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι ότι σε κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να πετύχουμε, να το πετύχουμε. Στην Οσετία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί υπάρχει παράλληλα και η αποσταλή του ΟΑΣΕ, και ερχόμαστε σε επαφή με Ρώσους, Γεωργιανούς και Νότιους Οσέτες, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτές τις συναντήσεις. Έχουν διαμορφώσει ένα επιχειρηματολόγιο θα έλεγα, το οποίο δεν τους δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και αυτό οφείλεται στην εξαφάνιση τριών ομάδων που εξαφανίστηκαν από πλευράς της διοικητικής γραμμής μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και οι Οσετιανοί πιστεύουν ότι οι Γεωργιανοί ξέρουν πολύ περισσότερα από όσα λέγουν και θεωρούν ότι για να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να πάρουν συμπληρωματικές πληροφορίες από τους Γεωργιανούς, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Έγινε όμως προσπάθεια, υπήρξε μια φάνταστη μορφή βοήθειας από τον αρμόδιο επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης ο οποίος προσέλαβε δύο ιδιαίτερα ε, ικανούς ερευνητές και οι οποίοι απλά βρήκαν αυτά τα οποία γνωρίζαμε για την υπόθεση αυτή. Και ο τελευταίος από αυτούς που έχει μείνει τώρα ολοκληρώνει την προσπάθειά του, αλλά φοβάμαι ότι αυτό δεν θα πείσει τους οσέτες να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ένα άλλο συστατικό θα έλεγα αυτών των μηχανισμών, ίσως το πιο σημαντικό, είναι η λεγόμενη θερμή γραμμή. Είναι ένα δίκτυο κινητών τηλεφώνων και στις δύο πλευρές και στους Οσέτες και στους κατοίκους της Απχαζίας και στους Γεωργιανούς και στους Ρώσους. Όταν υπάρχει ένα συμβάν, μέσα από αυτήν τη θερμή γραμμή, το δίκτυο αυτό, ανταλλάσσονται ιδέες για το τι έγινε. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μπορεί ο καθένας από πλευράς δικής του να δει πώς μπορεί να ελέγξει κάποιες ε, συνέπειες διεύρυνσης του προβλήματος. Αυτό λοιπόν είναι ένα μέσο το οποίο νομίζω ότι λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την φυσική συνάντηση των συμμετεχόντων, εμπλεκομένων μάλλον σε αυτή τη σύγκρουση σαν μια ενδιάμεση λύση. Συναντώμεθα τακτικά και με τους εκπροσώπους των συνοριακών φρουρών της Ρωσίας. Ενημερώνουμε τους Γεωργιανούς για τις συναντήσεις αυτές πριν και μετά. Και οι συναντήσεις αυτές έχουν αποδειχθεί θα έλεγα σχετικά παραγωγικές. Κλείνοντας, έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο στον τομέα της σταθεροποίησης, αν και τίποτα όπως είπα δεν είναι δεδομένο η συνέχιση της παρουσίας της αποστολής στην περιοχή είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Δεύτερον, κάναμε λιγότερη πρόοδο, σημειώσαμε λιγότερη πρόοδο στον τομέα της εξομάλυνσης της κατάστασης, έχουμε κάποια πρώτα βήματα θετικά στον τομέα της ελευθερίας διακίνησης, έχουμε επηρεάσει θετικά την ενδιάμεση λεγόμενη στρατηγική των Γεωργιανών, έχουμε κάνει μικρή πρόοδο στον τομέα της οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, αλλά απαιτούνται δύο για να χορέψει κανείς και ε, θέλει χρόνο για να πείσουμε και τις δύο πλευρές οι οποίες πολεμούσαν η μία την άλλη πριν δύο χρόνια να εμπλακούν με παραγωγικό τρόπο σε ένα τέτοιο μηχανισμό, κλείνοντας για τρίτη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχουν προσωπικό για την αποστολή μας. Είμαστε πολύ τυχεροί Έχουμε καλύψει το οργανόγραμμά μας κατά 100%. Βέβαια η οικονομική κρίση έχει αφήσει, αρχίσει να αφήνει ίχνη. Δεν είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη έκκληση για συνεισφορές από πλευρά κρατών μελών θα, απεδώσει, θα αποδώσει τα αναμενόμενα σε επίπεδο παρατηρητών. Θα ήθελα να μεταφέρετε λοιπόν στις κυβερνήσεις σας την ανησυχία μας αυτή ε, να τους πείσετε ότι η δουλειά που κάνουμε είναι θετική, είναι χρήσιμη και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεισφέρει. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Πρωτού να δώσω το λόγο στον κύριο Λιζέκ, τον Αντιπρόεδρο και εισηγητή ε, για τη Γεωργία, ένα ερώτημα. Το συμπέρασμά σας με φαίνεται σε αυτό το ερώτημα. Μιλήσατε για στελέχη, για προσωπικό πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βελτιώσετε στην αποστολή σας και τον εξοπλισμό τεχνικό, διοικητικής μέρημνας κτλ. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν αναφέρεται ε, στις αποστολές που ακούμε εδώ. Και είναι καλό να γνωρίζουμε ε, εάν υπάρχουν οι εξοπλισμοί σε ένα χώρο ο είναι δύσκολος. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη για τις λεπτομερείς πληροφορίες που μας έδωσε. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της κατάστασης. Σας παρακολούθησα και αν κατάλαβα υπάρχει μια νότα αισιοδοξία στα λόγια σας. Οπωσδήποτε η υποεπιτροπή μας αυτό το κοινοβούλιο θα υποστηρίξει στο μέτρο του δυνατού ε, την αποστολή σας και τις σχετικές επιχειρήσεις. Αλλά θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Ε, θα μεταβούμε στη Γεωργία και πιστεύετε κύριε Πρέσβη ότι θα μπορέσουμε να μεταβούμε στα κατεχόμενα εδάφη. Από ό,τι μας είπατε, αυτό μάλλον είναι αδύνατο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παρακαλώ επίσης ε, να μου πείτε αν υπάρχει ένα θετικό σενάριο διότι πρέπει κανείς να σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα θετικό σενάριο. Λοιπόν, το ερώτημά μου, η αποστολή μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ένα θετικό σενάριο, μια θετική εξέλιξη. Αυτό είναι το ερώτημα. θα υπάρξει συμφωνία νομίζω για την παρουσία ε, της αποστολής μας στην Νότια Οσετία και στην Απχαζία. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Εάν όχι, σε ποιο μέτρο αυτή η αποστολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να λειτουργήσουμε εάν συναυθεί συμφωνία με όλα αυτά τα μέρη για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια επιτυχημένη αποστολή σε αυτά τα εδάφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον ε, πρέσβη Χάμπερ για την ε, πολύ λεπτομερή παρουσίαση που μας έκανε. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Το πρώτο ίσως να είναι έτσι γενικό. Σε μια ακρόαση στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πριν από λίγες μέρες, ο Νταν Χάμιλτον από την ε, Ουάσιγκτον σχετικά με μια γενική παρατήρηση ότι δηλαδή καμιά φορά οι διάφοροι πυλώνες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντί, αντίκεινται ο ένας τον άλλον, είπε ότι δεν είναι απολύτως κατανοητό γιατί σε αυτή την περίπτωση με την αποστολή παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γεωργία. Ε, δεν έγινε αυτό στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Ερώτημα λοιπόν προς εσάς. Συγκεκριμένα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της αποστολής σε σχέση με μια πιθανή αποστολή του ΟΑΣΕ, αν μπορείτε να το συγκρίνετε. Δεύτερον, ένα ερώτημα σχετικό με τη νέα εντολή. Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό, δεν είναι κρυφό, ότι από τη μία υπάρχουν φωνές που θέλουν να ενισχύσουν την εντολή και από την άλλη υπάρχουν φωνές που θέλουν να αποδυναμώσουν, να μειώσουν λίγο την ισχύ της εντολής. και σχετικά με το ότι μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα δημιουργίας εμπιστοσύνη. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα και θέλω να μου πείτε εσείς τη δική σας ανάλυση. Ε, βλέπετε τη δυνατότητα ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην, αυτή, αυτή η, έμφαση στην, ε, στην ε, εμπιστοσύνη θα μπορούσε ίσως να βελτιώσει την πρόσβαση ας πούμε προς περιοχές της Νότιας Οσετίας της Απχαζίας. Θα ήταν ε, χρήσιμη η δική σας γνώμη. Τρίτον, για την επόμενη φάση. Πώς θα μετρήσετε την επιτυχία, το κατά πόσο η αποστολή είναι επιτυχής ή όχι. Η πρόσβαση, ας πούμε, είναι μέτρο επιτυχίας. Επίσης, κάποιοι εσωτερικώς εκτοπισμένοι που μπορούν ας πούμε να, να γυρίσουν πίσω στην, στην περιοχή τους αποτελεί σημείο επιτυχίας για σας. Ε, το να υπάρξει απόσταση από τα σύνορα είναι μέτρο. Το παράνομο, το παράνομο σημείο διέλευσης και η απόσταση από αυτό θα είναι σημείο επιτυχίας για σας πώς, πώς θα μετρήσετε την μελλοντική επιτυχία της αποστολής. Και τελευταία ερώτηση. Η ε, δουλειά που κάνετε δυσκολεύει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στο παρελθόν δεν είχε μία συγκεκριμένη σαφή ενιαία θέση σε ό,τι αφορά την παραβίαση ε, εναντίον της Ρωσίας. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε και, από, και εσείς και ο κύριος Κλόπενχάουερ κατά την άποψή σας τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε μια πιο συνεκτική και πιο σαφή θέση έναντι της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Νικολάη. Ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήματα σε σχέση με την αποστολή σας στη Γεωργία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν η μοναδική ευκαιρία για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Εξετίμησα πολύ την παρουσία σας εκεί και νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει, θα μπορούσε να ενισχυθεί η εντολή, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Πράγμα το οποίο οι πάντες επιθυμούν τι πιστεύετε για το νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί. Γιατί νομίζω ότι ο πρόεδρος Μετβέντεφ ενδιαφέρεται πολύ στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της άμυνας και στο στρατιωτικό τομέα. Μπορούμε ε, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και να περιλάβουμε και το φάκελο, το θέμα της γεωργίας. Μπορούμε, αν θέλετε, να ασκήσουμε κάποια πίεση και το δεύτερο ερώτημα αφορά τα θέματα της διοικητικής μέρημνας. Νομίζω ότι η διοικητική μέρημνα που χρησιμοποιείται στη Γεωργία δεν αρκεί και ίσως χρειάζονται περισσότερα για να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αποστολής. Αυτό είναι πιο σημαντικό για μας για να υπάρχει διαφάνεια, αξιοπιστία, ε, της Ένωσης, αλλά ώστε η αποστολή αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ η κυρία Λόζιν. Ναι, Πρόεδρε, σε σχέση και με την ε, προηγούμενη ανταλλαγή α, απόψεων, είχα κάποια ερωτήματα για, το, για τη δική σας ε, άποψη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. πρέπει να πω ότι η παρουσίαση του προηγούμενου προσκεκλημένου μου φάνηκε πολύ μονομερής. Και οι αναλύσεις που έκανε για τις διενέξεις, έτσι όπως τις παρουσίασε, μου φάνηκαν μονομερές. Ε, είπατε κάποια στιγμή εσείς ότι ο Υπουργό Ιστορικών της Γεωργίας έχει τελείως διαφορετική άποψη για την ασφάλεια ή ότι εν μέρη δεν υπάρχει διάθεση να υπάρξει συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, ε, ρωτώ, αναρωτιέμαι, προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανατολική ε, διάσταση της πολιτικής γειτονίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς ποια κατεύθυνση θα πάμε ε, σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά ζητήματα. Δηλαδή, οι επαφές θα εντατικοποιηθούν με τη Γεωργία. Και άλλο ερώτημα έτσι όπως ε, έχει τα, η κατάσταση και με την ε, Ουκρανία και η συμμετοχή της ε, Γεωργίας είναι πιθανή σε μια τέτοια ομάδα. Επίσης, συνεργασία για, για το περιθώριο χειρισμών υπάρχει και επίσης εγώ ανησυχώ με όλα αυτά που έχω ακούσει σήμερα και για την ε, εντολή της ε, κοινή ε, δράσης για το 376. Εκεί αναφέρεται ότι η αποστολή θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των υποδομών, των εγκαταστάσεων της, του τομέα της ενέργειας και των μεταφορών. Ερώτημα. Σε σχέση με αυτό, συγκεκριμένα, τι έχει γίνει. Ευχαριστώ. President. Sincere thanks for... Ονομάζομαι Τάτουνε από τη Λιθουανία με δύο μικρά ερωτήματα. Με ποιο τρόπο συγκεκριμένα η, ο βασικός πρωταγωνιστής η Ρωσία σέβεται την εντολή της αποστολής παρακολούθησης UMM. και παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι προβλέπετε για την εποχή μετά την ολοκλήρωση της αποστολής ε, παρακολούθησης. Τι θα συμβεί μετά. Thank you, uh, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη και κύριε Κόπενχάουρ, σε συνέχεια ε, των όσων είπε ο συνάδελφος, θα ήθελα ε, να μιλήσω για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη και την ελεύθερη διακίνηση. Τώρα, για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, Είπατε ότι προσπαθείτε να έχετε επαφές ε, με την κοινωνία των πολιτών εκατέρωθεν. Αυτό δεν λειτουργεί, είπατε, προς το παρόν. Τι μέτρα προβλέπετε, τι ιδέες προβλέπετε, σχεδιάζετε ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου ε, της για τον Νότιο Κάφκασο ε, έχουν ε, επισκεφθεί την περιοχή πριν από το Πάσχα και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να υποστηρίξουμε αυτές τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα για την ελεύθερη διακίνηση. Είπατε ότι προσπαθείτε άτομα τα οποία έζησαν στην περιοχή από τις δύο πλευρές ε, αυτών των διοικητικών ε, συνόρων να διακινούνται πιο ελεύθερα. Όταν όμως εμείς επισκεφθήκαμε αυτή την διοικητή γραμμή πριν από το Πάσχα, από την αποστολή ε, των ΗΕ, ορισμένοι μας είπαν ότι προσπάθησαν να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα για το τι μπορεί κανείς να κάνει προγράμματα, projects που θα έδιναν μεγαλύτερη πρόσβαση στα άτομα εκατέρωθεν αυτής δηλαδή, της διοικητικής γραμμής, δηλαδή προς βορρά και προς νότον της διοικητικής γραμμής. Έχει γίνει καθόλου πρόοδος σε αυτά τα προγράμματα, διότι μας είπαν ότι έτσι κι αλλιώ ορισμένοι περνάνε τα σύνορα από τη μία πλευρά ή την άλλη το βράδυ, όταν δεν τους βλέπουν οι φύλακες ε, των συνόρων. Υπάρχει πρόοδο σχετικά με την ελευθερία διακίνησης. Κάτι άλλο το οποίο ρώτησαν και άλλα μέλη της Επιτροπής. Η Γεωργία ζητάει μια εκτελεστική εντολή. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται ή σκοπεύετε να περιορίσετε την αποστολή. Νομίζω ότι η αποστολή πρέπει να παραμείνει, να επεκταθεί ακόμα. Και με μια διοικητική, για τη διοικητική εντολή δεν συμφωνώ προσωπικά. Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά. Και μια τελευταία παρατήρηση. Στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, για ε, την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, είχαμε διατυπώσει την ανησυχία μας, την απογοήτευσή μας σχετικά με την ε, απόφαση που εξήγηλε η ρωσική πλευρά να δημιουργηθεί ε, μια, μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ Νότιας Οσετίας και ε, Γεωργίας. Αυτό μας προβληματίζει, διότι αυτό σημαίνει ότι αυτές οι διοικητικές διαχωριστικές γραμμές θα γίνουν μόνιμες που δεν έχουν γίνει δεκτές διεθνώς. Ε, πώς θα αντιδράσετε, σκοπεύετε να αντιδράσετε και... Κύριε Πρόεδρε, εφόσον έχω το λόγο, θα ήθελα να κάνω και άλλη μια παρατήρηση η οποία ίσως έχει σχέση και με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Θα ήθελα να στραφώ στα μέλη της Επιτροπής αυτής και να ζητήσω την υποστήριξή τους σχετικά με θυλακούς ε, που έχουν σχέση με τη Ρωσία και τη Γεωργία. Ε, αυτή η σύμβαση η οποία υπάρχει θα αρχίσει να ισχύει, να ισχύει την 1η Αυγούστου αλλά υπάρχουν και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπογράψει, επικυρώσει αυτή τη σύμβαση. Υπάρχει μια πρωτοβουλία από την κοινωνία των πολιτών που ε, θα υποβάλουν ένα προφορικό ερώτημα στο Στρασβούργο την επόμενη φορά με ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία ε, το γνωρίζουν, να, να ζητήσουν α, την υποστήριξη όλων των ομάδων σε, αυτό, σε αυτή την προφορική ερώτηση που θα γίνει ε, στο Στρασβούργο την επόμενη φορά. Ο κύριος Στάθμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, κύριε Πρέσβη, και συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε εκεί, διότι και ο προηγούμενος ομιλητής εδώ μας είπε ότι υπάρχει μια κλιμάκωση ορισμένων πραγμάτων μετά τον Αύγουστο. Και με τα γεγονότα που παρουσιάσατε φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Επίσης, ε, είπατε ότι κερδίσατε την καρδιά των ανθρώπων. Και αυτό το έντυπο το δείχνει. Και είναι σημαντικό σε οποιαδήποτε αποστολή, στρατιωτική ή μη στρατιωτική, να συμφωνεί ο λαός. Από αυτή την άποψη όμως θα ήθελα να σας κάνω το εξή ερώτημα επειδή ασχολείστε με τους ανθρώπους εκεί, με τους απλούς ανθρώπους και από τις δύο πλευρές της γραμμής, των, ε, της επικίνδυνης γραμμής. Ποιο είναι το συνέστημα των ανθρώπων εκεί, τι θέλουν. Πιστεύετε ότι βαίνουμε προς μια κατάσταση τύπου Κωσυφοπεδίου ή Κύπρου ή υπάρχει ακόμα μια ελπίδα για επανένωση της Γεωργίας στο άμεσο μέλλον ελπίζουμε τελευταία παρέμβαση, ο κύριος Ερενάουζερ. Ευχαριστώ. Η ποιότητα των πολιτικών αποφάσεων πάντα εξαρτάται και από τις πληροφορίες που λαμβάνει κανείς. Μιλήσατε για το ότι οι πολιτικές αποφάσεις και αυτοί που τις αναλαμβάνουν μόνο γενικώ είναι ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες που έχουν. Ερώτημα τεχνικό λοιπόν πώς λειτουργούν οι γραμμές της, ε, των γνωμοδοτήσεων, δηλαδή σε ποιον δίνει αναφορά κάποιος μια ομάδα παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πληροφορίες από εθνικό επίπεδο πώς λαμβάνονται. Και ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Merci, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Κλάπενάουρ, κύριε Άμπερ, σας αφήνω να απαντήσετε ανάλογα με τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι, πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού βεβαίω, αλλά δεν μπορώ να ξεπεράσω τα πλαίσια της εντολής μου που δεν είναι πολιτική. Αλλά, όπως γνωρίζετε, εκτελώ ε, εντολή, αποστολή μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο και βεβαίως στο μέτρο του δυνατού. Τώρα, το πολιτικό πλαίσιο που έχει δοθεί ε, καθορίζεται από την συμφωνία μεταξύ των δύο προέδρων μετά από τον πόλεμο. Ε, το πρώτο μας αντικείμενο, όπως είπε ο κ. Πρέντης, ήταν να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και κατόπιν να προχωρήσουμε σε ομαλοποίηση της κατάστασης και ε, σε μετρεκοδόμηση εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει πολιτική εντολή, να αναφερθούμε στο status quo ex ante και δεν μπορούμε να πιέσουμε την κατάσταση. Δεν μπορούμε να πιέσουμε την κατάσταση. Καμία κατάσταση. Πρόκειται για, μια μη στρατιωτική αποστολή, όχι στρατιωτική αποστολή, το οποίο δείχνει και την περιορισμένη φύση ε, των, της εντολής μας. Συνεπώς το θέμα να επανέλθει αυτή η αποστολή στις ε, περιοχές de facto, ουσιαστικά είναι πολιτικό θέμα. Ε, αν ε, μετρήσουμε την επιτυχία της αποστολής, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να μετρήσετε ε, την αποστολή σε σχέση με την Νότια Οσετία και τη Ρωσία, διότι τότε γίνεται πολιτικό θέμα. Αλλά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και την ομαλοποίηση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Η φιλοσοφία βεβαίω, όπως είπε ο κύριος Πρέσβη, είναι τα... Ε, να μην υπάρχουν αυτά τα σύνορα, να χαλαρώσει τα σύνορα και να υπάρξει απεμπλοκή τη κατάσταση. να υπάρχει επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή είναι η βασική μας φιλοσοφία. Θα ήθελα να επανέλθω πάλι στο ιστορικό γιατί δεν είμαστε ο ΑΣΕ. Αυτό, όπως σας είπα, ε, τότε ήταν πολιτική αποστολή εμείς. Θα ε, Είμαστε διαδεμένοι να συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ και τον ΑΣΕ και συνεργαζόμαστε. Αλλά αυτή ήταν μια πολιτική απόφαση από τους εμπλεκόμενους ε, στην διένεξη και λυπούμεθα που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά εφόσον αυτή ήταν η πολιτική απόφαση. Δεν τους διώξαμε εμείς. Και σεβόμαστε πολύ το έργο το οποίο επιτέλεσε ο ΑΣΕ εκεί. Έστω ότι η πολιτική κατάσταση μας επιτρέψει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο από την άλλη πλευρά της διοικητικής γραμμής τότε θα άλλαζε η εντολή μας. Θεωρητικά νομίζω όχι. Ίσως αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσει από πλευράς προσωπικού, θα μπορούσαμε να κάνουμε ήδη ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό εξαρτάται από τα καθήκοντα που θα μας ανατεθούν σε μια νέα κατάσταση και κατά πόσο θα πρέπει να, αν θα αλλάξει εντολή και αν θα αλλάξει ο αριθμός ε, των ατόμων που μας βοηθούν. Θα σταματήσω εδώ και είμαι βέβαιο ότι ο κύριος Πρέσβης θα καλύψει τα υπόλοιπα ερωτήματα. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, το θέμα του εξοπλισμού. Επιχειρούμε για μία διετία και έχουμε αρκετά από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε πλέον. Βέβαια μας πήρε χρόνος για να τα έχουμε σε επίπεδο εξοπλισμού μας έχει βοηθήσει το CPCC και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση έτσι ώστε ο εξοπλισμός να μπορεί να είναι στη διάθεσή μας, στη διάθεση της αποστολής γρηγορότερα. στην αρχή ήμασταν εκεί με τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ και έβλεπε κανείς ότι αυτές οι δύο οργανώσεις έχουν μεγαλύτερη ιστορία και μεγαλύτερη εμπειρία στη συγκεκριμένη στο συγκεκριμένο πεδίο ειρηνευτικές ε, πολιτικές παρεμβάσεις, μη στρατιωτικές μάλλον παρεμβάσεις. Και έχουν πολύ γρηγορότερες διαδικασίες από εμά και πολλά έχουμε να μάθουμε από αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ήθελα να μειώσω ε, σε καμία περίπτωση το πόσο υπόλογοι παραμένουμε οικονομικά. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει να μην φύγει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό μας με γρηγορότερες προμήθειες υλικού. Χρειάστηκε 1,5 χρόνο να φτάσουμε εκεί που θα έπρεπε να ήμασταν από την αρχή. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να επιταχύνουμε σε σχέση με τον ΟΙΕ και τον ΟΑΣΕ. Για την ερώτηση Λίζεκ αν πάει κανείς τα κατεχόμενα. Ναι, αν ζητήσει κανείς ε, ε, την άδεια των αρχών ε, θα το κάνουν, αλλά στην ουσία θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για αναγνώριση της δικής τους εκεί παραμονής και το αποφεύγουμε. η αποστολή είναι διατεθειμένη, πιστεύει μάλλον ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Ναι, το πιστεύουμε αυτό σε σχέση με τις de facto οντότητες τις εθνοτικές που υπάρχουν. Πιστεύω ότι η εντολή μας η οποία ισχύει για το σύνολο του εδάφους της Γεωργίας μπορεί να παίξει θετικό ρόλο. Αυτή τη φάση βρισκόμαστε μόνο στην νότια πλευρά της διαχωριστικής γραμμής. Έχουμε πετύχει περισσότερα από ότι ο ΑΣΕ και τα Ηνωμένα Έθνη είχαν πετύχει τη στιγμή τουλάχιστον που πήγαμε εμεί εκεί και αυτό προσδίδει ε, στον πληθυσμό της περιοχής και από τις δύο πλευρές της ε, διαχωριστικής γραμμής μια κάποια ασφάλεια και μας το έχουν πει αυτό. Ακόμα και αν μας δίνεται η δυνατότητα όμως να πάμε στην Νότια Ασετία και την Απχασία, αυτό θα το κάνουμε παραμένοντας ορατή θα έλεγα και από τις δύο πλευρές. Μετά τέθηκε το ερώτημα Κόφερ για την επόμενη εντολή. Αύξηση ή μείωση. Νομίζω ότι μπορούμε να παραμείνουμε ως έχουμε. η δύναμή μας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και να αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες που έχουμε εμείς στις de facto ανεξαρτητοποιημένες περιοχές. Γι' αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν τη δύναμη που έχουμε. Δεύτερον, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Ο βασικός πυρήνας της αποστολής αλλάζει η ενέργειά μας πηγαίνει περισσότερο στο θέμα της ελευθερίας διακίνησης των πληθυσμών, αλλά μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές αποστολές αργότερα. Πάντως, προς στιγμή, η μείωση των μελών της αποστολής θα ερμηνευτεί αρνητικά και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, ή από όλες μάλλον τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν υπάρξει παράταση ή όχι. Είμαι λοιπόν, έχω αμφιβολίες. Η λογική της ρησικής πολιτικής σε σχέση με τον ΟΑΣΕ και τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι οι αποστολές που ήταν παρούσες και από τις δύο πλευρές της διαφορετικής γραμμής δεν θα έπρεπε να παραταθεί η διάρκεια τους. Εμείς έχουμε εντολή για το σύνολο του εδάφους της Γεωργίας, αλλά δεν ήμασταν εκεί εξ αρχής. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφορετική συνθήκη. Πώς λοιπόν μπορούμε να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας μας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όταν εμείς πήγαμε εκεί, τις πρώτες εβδομάδες και μήνες της αποστολής, δεν μπορούσα να βγω από μία συνάντηση χωρίς να με ρωτήσει ένας δημοσιογράφος γεωργιανός πότε θα μπορέσετε να μπείτε στην Οσετία και την Αφχαζία. Το ερώτημα δεν μου τίθεται όμως τώρα πια πλέον. Γιατί οι Γεωργιανοί συνειδητοποιούν, θα έλεγα, την αξία της πολιτικής μη αναγνώρισης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για αυτούς εν πολύ αντικαθιστά, θα έλεγα, τη δυνατότητα πρόσβασης. Για την κοιλάδα του Αχαλγούρη. Εκεί εξαρτώνται τα πράγματα από την επιθυμία των νότιων οσετών, δηλαδή να επιτρέψουν το ελεύθερο πέρασμα πληθυσμού και ε, αγαθών. Το αχαγκούρι είναι για αυτούς θα έλεγα ένα υπόδειγμα εθνοτικής συμφιλίωσης και συμβίωσης που δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές. Έχουν λοιπόν κάθε λόγο και οι οσέτες να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Και μπορεί πάντως να βελτιωθεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Σε άλλες περιοχές, περιοχή Πέρβη, έχει υπάρξει μια κάποια πρόοδος. Είναι η μοναδική περιοχή εκτός Νότιας Οσετίας, την οποία εξακολουθεί να κατέχει η Ρωσία υπάρχουν και δίδονται διαφορετικές ερμηνείες αυτής της κατάστασης, αλλά αυτό είναι σαφές και οι Ρώσοι συμφωνούν μαζί μας και έχουν εκφράσει την πρόθεση να ε, αποχωρήσουν από την περιοχή αυτή. Αυτή στιγμή βέβαια ε, δημιουργηθεί μια συνδετήρια οδός. για την κυρία Νικολάη. Τα της επιμελητίας έχω ήδη δώσει απαντήσεις. Λούσινγκ. για τις διαφορετικές εκτιμήσεις ανάμεσα σε μας και το Υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας. Το Υπουργείο λέγει ότι αυτοί οι οποίοι μένουν εκεί κοντά στην περιοχή αυτή της διαφορετικής διαχωριστικής γραμμής πυροβολούν στον αέρα και κανείς δεν τραυματίζεται, αλλά παρόλα αυτά οι εκφοβιστικές αυτές πρακτικές κάνουν τον κόσμο να μην θέλει να μένει εκεί. Και γι' αυτό το Υπουργείο λέει ότι για αυτούς που μένουν στη γραμμή για να νιώθουν προστατευμένοι θα πρέπει να έχουμε μια μαζική στρατιωτική παρουσία. Εμείς λέμε ότι δεν θα πρέπει να ασκεί κάτι τέτοιο, γιατί η μικρότερη παρουσία στρατιωτική, ορατή, θα μειώσει τις εντάσεις και έμεσα θα δώσει μια αίσθηση ασφάλειας στον τοπικό πληθυσμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα μιας μορφής συνεργασίας με την άλλη πλευρά και ιδιαίτερα τους Ρώσους συνοριοφύλακες, γιατί οι κάτοικοι της Αφγαζίας και της Νότιας Οσετίας στην ουσία έχουν εκχωρήσει την επίβλεψη των διαχωριστικών γραμμών τους στην ρωσική συνοριοφυλακή. Για συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ δεν έχω εντολή γύρω από αυτό. Υπήρξε το θέμα της ενέργειας το σφράγμα Ινγκούρι δίδεται σαν παράδειγμα, θα έλεγα, για τους περιορισμούς στην συνεργασία που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε αντιτιθέμενες ομάδες. Ελέγχεται εδαφικά από την Τυφλίδα, αλλά παρόλα αυτά η περιοχή, ε, η μονάδα αυτή ελέγχεται από την Νότια Οσετία. Και γι' αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να δουλεύει η μονάδα αυτή είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας, επιβεβλημένη συνεργασίας, η οποία δυστυχώς όμως δεν φαίνεται να δημιουργεί αντίστοιχες καταστάσεις. Δεν έχει λειτουργήσει παραδειγματικά. Για τον κύριο Λάντσμπεργκης. Μετά το τέλος της εντολής, τι θα γίνει. Κάποια στιγμή θα τερματιστεί η εντολή. Το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και θα θέλαμε η κατάσταση που θα αφήσουμε πίσω να είναι διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα. Αν η ρωσική στρατηγική αποδώσει, θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, ότι σε κάποια φάση δεν θα υπάρχει ανάγκη για κάποια κομμάτια της αποστολής αυτής. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Γεωργίας η στρατηγική αυτή τουλάχιστον να πετύχει ιδιαίτερα στον τομέα της ελευθερίας διακίνησης. Γιατί εκεί νομίζω ότι με τη συλλογική εμπειρία την οποία έχουμε σαν αποστολή μπορούμε τα πράγματα να τα βελτιώσουμε. αν γίνεται σεβαστή η εντολή της αποστολής μας. Ναι. Οι Γεωργιανοί, δεν ξέρω αν σας είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γεωργίας, οι Γεωργιανοί θέλουν να μετατρέψουν την αποστολή μας σε μια ένοπλη αποστολή α, ε, τήρησης ειρηνευτική. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Δεν συνειδητοποιούν όμω ίσω οι Γεωργιανοί ότι αυτό προποθέτει ένα εντελώ διαφορετικό περιβάλλον. Μια τέτοια ειρηνευτική δύναμη θα είναι μια δύναμη διαμεσολάβηση, αλλά προς τον παρόν όπως μας έχουν πει είναι σχετικά ικανοποιημένοι με την κατάσταση ως έχει και πιστεύουν ότι η αποστολή μας λειτουργεί θετικά για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη συνοριακή γραμμή. Λούνατσεκ για την κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώ, δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα από όσα είπατε. Υπάρχουν αρκετέ πρωτοβουλίε από διεθνείς ΜΚΟ έτσι ώστε άμαχοι και από τις δύο πλευρές να έρθουν σε επαφή. Έγινε μια πρώτη επαφή στην Κωνσταντινούπολη πριν λίγες εβδομάδες, πήραμε μέρος έτσι ώστε να σημειώσουμε την επαφή αυτή, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και επαφές. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες το σύστημα των κινητών τηλεφώνων της Γεωργίας δεν λειτουργεί στην Οσετία και απαιτείται πολύ υπομονετική προσπάθεια εφόσον μπορείτε να μας βοηθήσετε με τις επαφές που έχετε με μη κυβερνητικές οργανώσεις από την άλλη πλευρά, αυτό θα ήταν καλό. Λόγω της εικόνας που έχει αυτή τη στιγμή η αποστολή μας δεν είμαστε σε θέση να τα εξηγήσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά της μεθοριακής γραμμής. Έχουμε συναντήσει και κάποιους δημοσιογράφους από τις περιοχές ε, ε, ε, που έχουν αποσκυρτήσει αλλά προς το παρόν οι επαφές βρίσκονται σε ένα πρόωρο στάδιο. οι αναφορές τις οποίες κάνουν ε, οι παρατηρητές. Οι παρατηρητές είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον άμαχο πληθυσμό, με την αστυνομική, αστυνομία, συλλέγουν πληροφορίες και οι πληροφορίες αυτές μετατρέπονται σε εκθέσεις από τους υπεύθυνου αξιωματικούς προς το στρατηγείο και το στρατηγείο συνδυάζει τις εκθέσεις αυτές και σε εβδομαδιαία βάση, μηνιαία βάση και εξαμηνιαία βάση εκδίδει ειδικέ εκθέσεις ή θεματικές εκθέσεις. Σε τομείς όπου σαν παράδειγμα άρδευση κατά μήκο της μεθοριακής γραμμής ή επαφές με μικιό. Χρήση των γεωργικών γεών Αυτά είναι θέματα τα οποία προβλέπονται και από το CPCC και από τη συνεργασία με τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ε, Για τον κύριο Στάτσνη. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι από τους πολίτες λένε ότι είχαμε και κάποιες διεθνείς ε, αποστολές τα τελευταία 20 χρόνια και δεν άλλαξαν τελικά την κατάσταση. Άλλοι λένε ε, είμαστε τόσο ευγνώμονες που είσαστε εδώ γιατί αισθανόμαστε ασφάλεια. Ειδικά με τα, το, τα τον Αύγουστο. Βέβαια η κοινωνία είναι γεωργικοί, δεν τους νοιάζουν τα πολιτικά, τους ενδιαφέρει να μπορούν να έχουν τις σοδιές φουντουκιών που είχαν, να μπορούν να κάνουν τη ζωή που είχαν. Υπάρχει δηλαδή με αρκετά παθητική στάση από τους πολίτες, αλλά εμένα πάντα με εκπλήσει μετά από δύο χρόνια υποτέπου παρουσίας πόσο συχνά έχουμε θετικές ε, απόψεις. Στατικές απαντήσει γιατί τελικά όντω προσπαθούμε να βοηθήσουμε να μάθει ο κόσμος τι είμαστε και τι κάνουμε εκεί και γιατί. Και κάνουμε έτσι αρκετά, έχουμε αρκετά προγράμματα που προσπαθούν να φτάσουν σε όλου του πολίτε και τελικά αποδίδουν. Αυτά νομίζω. The FSB border guards. Well, yes, the FSB border guards. As I said, um... Για του συνοριοφύλακε. Όπω είπα, για την ασφάλεια της γραμμή, γραμμής, ε, τα αποτελέσματα είναι θετικά. Από τη μία, όπως ξέρετε, συμμορφούμενοι και με την νομική άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα να είμαστε εκεί. Απ' την άλλη πρέπει να συνεργαστούμε σε ένα βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε γίνονται κάποιες περιπολίες, αλλά ε, νομίζω ότι είναι αρκετά θετικά τα πράγματα. Τώρα, ο, οι συνοριοφύλακες ε, αποτελούν ε, την ε, αντίθεση στις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες συνήθως αναλαμβάνουν τα σύνορα και που συνήθως αφήνουν ε, ελεύθερα τα σύνορα για να περνούν οι πολίτες. Ε, ο στρατός όμως έκλεισε τα σύνορα όταν ανέλαβε. Η οργάνωση του διοικητικού, της διοικητικής συνολικής γραμμής που θα οδηγήσει. Θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα είναι πιο δύσκολο για τους πολίτες να περάσουν την διοικητική γραμμή και να πάνε στην άλλη μεριά ή θα ομαλοποιήσει τα πράγματα και θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και, νό και ομαλότητα. Γιατί ε, συνήθως ε, δωροδοκούσαν τους συνοφύλακες για να περάσουν απέναντι οι περισσότεροι. Και αυτό μειώνεται όλο και περισσότερο όταν, ε, όσο αναλαμβάνουν τα, την οργάνωση οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι χτίζουν διάφορες ε, εγκαταστάσεις για, τα, για τους συνοριοφύλακες τους. Οι υποδομές ε, είναι πραγματικά τεράστιες, είναι εντυπωσιακά τα κτίρια, δηλαδή μπορούμε να τα δούμε. Είμαστε κοντά βέβαια από την διοικητική γραμμή, αλλά μπορούμε να τα δούμε. Και για την Απχαζία, ξέρετε ότι ε, συνεργαζόμαστε και με το δορυφορικό κέντρο και λαμβάνουμε πληροφορίες και από αυτούς για το πώς είναι τα πράγματα εκεί. Και η απάντησή σας αυτό ποια είναι. Οπότε είναι σαν να προσπαθούν να, να καταστήσουν αυτό το σύνορο το πραγματικό σύνορο. Είπατε ναι, ωραία, έχετε καλέ επαφέ, αλλά όταν αυτοί δημιουργούν όλα αυτά τα τεράστια σύνορα, είναι σαν να θέλουν να καταστήσουν αυτό το νέο σύνορο και να αποτρέψουν οποιονδήποτε από το να περνά στην απέναντι όχθη. Εμεί είμαστε πολιτική αποστολή. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε με κάποιο τρόπο αυτό που κάνουν. Βεβαίω οι Ρώσοι και οι Απχάζοι και οι Οσέτοι ε, θεωρούν ότι αυτή η γραμμή είναι ένα σύνορο και θέλουν να φαίνεται και ο σύνορο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι απλώς να εξασφαλίσουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, και αυτό χρειάζεται ένα βαθμό συνεργασία, ότι η συνοριακή γραμμή θα είναι όσο το δυνατόν πιο διάτρητη για να μπορεί κανείς να περνά. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις κατάχρηση ή διαφθοράς τότε να του το γνωστοποιούμε, γιατί σε πολλέ περιπτώσεις δεν το ξέρουν καν. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θα βοηθήσει την στρατηγική της γεωργίας, θα βοηθήσει τις επαφές μεταξύ των πολιτισμών και στις δύο πλευρές, των πολιτών συγγνώμη και στις δύο πλευρές, οπότε θα ενισχύσει το στόχο της γεωργίας. Μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε στα όρια του εφικτού, του δυνατού μπορούμε να κινούμε τα πάντα. Κύριε κύριε ε, Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις που δώσατε. Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε για την υποδοχή που θα επιφυλάξετε στην κοινοβουλευτική μας αντιπροσωπεία τον Ιούλιο. Μετά από αυτή την επίσκεψη και ευκαιρία της έκθεσης για τη Γεωργία θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναβρεθούμε στις 12 Ιουλίου.